Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αυτή την κοινή ακρόαση με θέμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το πρώτο τμήμα αυτού του σεμιναρίου θα διεξαχθεί υπό την Προεδρία του Ρομπέρτο Γουαλτιέρη, που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Εγώ θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και θα προεδρεύσω στο δεύτερο τμήμα των εργασιών μας. Βρισκόμαστε στις παραμονές της έγκρισης ενός κανονισμού που θα παρατείνει και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πρόεδρου Γιούγκερ εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ανάληψη των καθηκόντων του. Προσπάθησε με το επενδυτικό αυτό σχέδιο να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό έλλειμμα που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάνω από 10 χρόνια πώς θα βοηθήσουμε τους επενδυτές, είτε είναι δημόσιοι, δημόσιοι φορείς, είτε ιδιωτικοί, ώστε να κινητοποιήσουν τα απαραίτητα κονδύλια για να καταστήσουν πιο στεναρές και εύρωστες τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πριν λοιπόν την ε, παράταση, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΕΦΣΙ θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανταπεξήλθε στην αποστολή της με την απαραίτητη και δέουσα επιμέλεια. Η, η οικονομική κλάδη έλαβαν τις ε, απαραίτητες απαντήσεις που περίμεναν. Οι διάφορες ε, περιφέρειες, οι διάφοροι φορείς ε, που εποφελήθηκαν από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου του, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων πώς αξιοποίησαν αυτές τις δυνατότητες. Όλα αυτά θα εξετάσουμε σήμερα με τους εμπειρογνώμονές μας και τα διδάγματα που θα αντλήσουμε από το σημερινό σεμινάριο θα μας χρησιμεύσουν στις συζητήσεις του σχεδίου κανονισμού που όπως σας είπα στόχο έχει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και ίσως μεταφέρουμε το μοντέλο, το πρότυπο αυτό του Ταμείου σε, άλλα, σε άλλους τομείς, όπως στο θέμα της ε, αηφόρου ανάπτυξης στις γειτονικέ μας χώρες ή στις αφρικανικές χώρες. Του τουλεχθέντος θα δώσω το λόγο στον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη που θα προεδρεύσει, όπως σας είπα, γύρω στις εργασίες μέχρι τις 5-5.30 στο πρώτο τμήμα του σεμιναρίου. Ευχαριστώ Ζαν και σας ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο αυτό. Μάλιστα έχουμε απευθείας αναμετάδοση της ε, συνεδρίασής μας και από το διαδίκτυο, οπότε όσοι δεν έχουν θέση μπορούν να παρακολουθήσουν και εκτός αίθουσης ε, τις συζητήσεις. Βέβαια, αν προτιμάτε να είστε στην αίθουσα όρθιοι, πολύ ευχαρίστω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα, αφιέρωσε μεγάλη προσοχή, χρόνο, και προσπάθειες σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο που αποτελεί νευραλγική σημασία πρωτοβουλία και επιχειρεί την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη γεφύρωση του τεράστιου αυτού επενδυτικού ελλείμματος. Οπότε θα κάνουμε ένα απολογισμό το πρώτο χρόνο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα περιμένουμε τη σχετική έκθεση αξιολόγηση από το πρώτο ΕΦΣΙ και περιμένουμε και το ΕΦΣΙ 2 που πέραν της διεύρυνσης και της αύξησης ε, θα βελτιώσει το επενδυτικό αυτό σχέδιο. Γιατί λειτουργεί εύρυθμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ακόμη. Και μάλιστα ένα θέμα που είναι σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα της αγοράς, και να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο για καλύτερο συνδυασμό, ανάμιξη κονδυλίων ή για καλύτερη εφαρμογή σε ένα πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής επενδυτικής στρατηγικής. Οι επενδύσεις που καλύπτονται από τις εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να συνδυαστούν με αυτές άλλων επενδυτικών ταμείων. Ε, του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής και φυσικά θα εξαρτηθούν όλα και από την ικανότητά μας να προσελκύσουμε και να κινητοποιήσουμε συμπληρωματικές ε, επενδύσεις. Μίζον ζήτημα λοιπόν αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα συμβάλλετε στη συζήτηση. Πρώτα θα ακούσουμε τους δύο συνεισηγητές μας και από την εκτελεστική και από την νομοθετική έκθεση και θα ακούσουμε μετά τους καλεσμένους μας και μετά την παρουσίαση και των εμπειρογνωμόνων θα έχουμε ελπίζω καρποφόρα συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον, επιτρο... στον εισηγητή τη ΕΚΟΝ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στον Ούτο Μπούλμαν. Σα ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ και σένα, Ρομπέρτο. Αξιότιμοι καλεσμένοι, καλώ ήρθατε. Απευθύνω ιδιαίτερα εγκάρδιο χαιρετισμό στου εμπειρογνώμονέ μα. Χαίρομαι ιδιαίτερω που καταφέρατε και ήρθατε και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε τεράστια διακομματική πλειοψηφία υπέρ της σύστασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΦΣΥ. Και Συμφωνήσαμε και με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράτασή του και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του. Και συμφωνώ απόλυτα με τον συνεισηγητή, τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε, και με του άλλου και οδησηγητές με του οποίου είχαμε πολύ επικοδομητική συνεννόηση στο παρελθόν. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι θα θέλαμε περισσότερες και καλύτερες συμπληρωματικές επενδύσεις. Αλλά είμαστε και, είμαστε πολύ καλοί φίλοι με το ΕΦΣΥ, αλλά οι φίλοι δεν συμφωνούμε τα πάντα, ούτε λες όλα ναι. Οι φίλοι έχουν καθήκον να είναι και επικριτικοί και να υποδεικνύουν τις αδυναμίες εφόσον τις εντοπίζουν. Γι' αυτό και σήμερα θα κάνουμε έναν απολογισμό. Θα αναλύσουμε τα επιτεύγματα του ΕΦΣΥ, αλλά και θα δούμε τι επιδέχεται βελτιώσει στη δεύτερη φάση λειτουργίας του. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το έργο του, οι, οι συνομοθέτες το ίδιο με το πρώτο ΕΦΣΥ, γιατί επιτύχαμε πραγματική συμπληρωματικότητα και είχαμε ενδιάμεσες δομές πολύ στεναρές που ήταν απαραίτητες γιατί τα κράτη-μέλη ήταν απρόθυμα για άμεσες επενδύσεις στο νέο αυτό φορέα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης υπογραμμίσαμε την ανάγκη να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιμένουμε τώρα την σωστή και πλήρη εφαρμογή όλων των επιμέρους μέτρων ε, εγώ θα έλεγα ότι η εφαρμογή, η εκτέλεση έχει αποτελέσματα από ποσοτική άποψη που μπορεί βέβαια να μην είναι αρκετή τελικά για ολόκληρη την Ευρώπη αλλά ποσοτικά μέχρι στιγμής το ΕΦΣΙ έχει αποφέρει καρπούς. Τώρα δούμε την ποιότητα. Εκεί έχουμε κάποιες παρατηρήσεις να κάνουμε γιατί η προσθετικότητα είναι σημαντική, αλλά είδαμε και κάποια προγράμματα και σχέδια που θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί διαφορετικά, όχι από τον κοινοτικό προπολογισμό. Επίσης είχαμε και ένα πίνακα επιδόσεων. Αυτός ο πίνακας επιδόσεων είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός ε, για να ε, προβάλλουμε τα προγράμματα που χρειαζόμαστε πραγματικά για να κάνουμε πιο βιώσιμη την ευρωπαϊκή οικονομία, πιο μελλοντοστραφή και οι μελλοντικέ μας ε, προκλήσεις αφορούν και τη χρησιμότητα αυτού του πίνακα επιδόσεων. Επίσης, επενδυτικές πλατφόρμες. Είπαμε, ε, ναι, όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν καλές ιδέες και σχέδια θα πρέπει να δοκιμάσουν και αυτές την τύχη τους και να τύχουν κάποιε υποστήριξει. Μέχρι στιγμής μόνο λίγες επενδυτικές πλατφόρμες ε, δημιουργήθηκαν. Γιατί λοιπόν τόσο λίγες, πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Γεωγραφική πολυμορφία και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί έχουμε ιδιαίτερες ανάγκες και στην κεντρική Ευρώπη και στη νότια Ευρώπη. Έχουμε εξαντλήσει τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε πραγματικά αυτούς που χρειάζονταν συμπληρωματικές επενδύσεις. Διαφάνεια. Ναι, θέλουμε να γνωρίζουμε ε, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έχουμε κάποια προβλήματα ακόμη με την ιεραρχία του συστήματος λήψης αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει και με τον τρόπο διακυβέρνηση ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης, πρέπει να στηρίξουμε τις περιφέρειές μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, προσφυλές και στον συνεισηγητή Ζωζε Μανουέλ Φερνάντες. Επίσης έχουμε το θέμα του κόμβου παροχής επενδυτικών συμβουλών. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τις περιφέρειες και να προβάλλουμε καλύτερα το, τους μηχανισμούς του ΕΦΣΥ για να γίνουν πιο αποδεκτοί και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτά είναι μερικά από τα ε, ερωτήματα που θα θέσουμε στη δεύτερη φάση, μετά τον απολογισμό που θα κάνουμε της πρώτης φάσης και μετά θα δούμε τι νομοθετικές ρυθμίσεις θα προταθούν για το δεύτερο εύση, μετά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια των καλεσμένων εμπειρογνωμόνων μας και των συναδέλφων. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε, Ούντο. Και τώρα ο συνεισηγητής από πλευράς προϋπολογισμών, ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα μιλήσω πορτογαλικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Εμείς, εδώ και 1,5 χρόνο, αναρωτιόμασταν κατά πόσο αυτό το ταμείο θα ήταν πραγματικά λειτουργικό και κατά πόσο ο πολλαπλασιαστής ε, του 2015 δεν θα ήταν ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόσκομα. Ευτυχώς ε, φτάσαμε στο ύψος των προσδοκιών, ε, μπορέσαμε να ανοίξουμε διόδους για επενδύσεις και ως προς τις ε, ΜΜΕ και η δίωδος που αφορά τις επενδύσεις ήταν μέσα στις προσδοκίες. Ε, είχαμε 28 κράτη-μέλη και είχαμε, και είχαμε 68 δις ως επίπεδο επενδύσεων. Μπορούσαμε λοιπόν να βελτιώσουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να προβούμε και σε μια καλή ερμηνεία του κανονισμού. Ο, όπως είπε και ο Ούντο Μπούλμαν, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει ο προσθετικός παράγων και όταν υπάρξει θα πρέπει να ερμηνευτεί καλώς. Πρόκειται για ένα ανοιχτό ταμείο και θα πρέπει να δείξουμε ενεργή πολιτική έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και την εδαφική συνεκτικότητα. Ως προς τον κανονισμό θα πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερα μικρά σχέδια και προγράμματα από αυτά που υποστηρίζουμε. Δηλαδή, καταρχήν οι πλατφόρμες που δεν χρησιμοποίησαμε ούτε διασυνοριακά. στο τομέα της ενέργειας θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Και γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το Ταμείο ε, Εγγυήσεων μέσα στα πλαίσια ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Άρα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να υπάρξουν διευκρινήσεις και να γίνουν και επενδύσεις στη γεωργία, στον κοινωνικό τομέα, στον ε, τομέα της ε, αλίας και της ηχθειοκαλλιέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε αυτό το ταμείο με τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και τα διαρθρωτικά. Είχαμε 13 δις μέσα στα πλαίσια του 16 που δεν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως για τις ΜΜΕ, για, τις, για την νεότητα, για τα πανεπιστήμια, για την καινοτομία, για την τεχνολογία και την έρευνα. Και υπάρχουν και οι πλατφόρμες αυτές όπου μαζί με το ΕΦΣΥ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία. Να υπάρχει δηλαδή συμπληρωματικός χαρακτήρας. Αποζητούμε πληροφορίες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον κανονισμό. Όταν μιλώ για μικρά προγράμματα, ο κανονισμός δεν ορίζει ένα ελάχιστο όριο αλλά αν υπάρχουν προγράμματα κάτω από 50-25 εκατομμύρια, ε, δεν βρίσκουν σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλο όμως 50 εκατομμύρια στο Βερολίνο και άλλο 50 εκατομμύρια στη Λισαβόνα ή σε ορισμένες απομακρυσμένες περιφέρειες της ε, Γερμανίας. Και αυτό αφορά και το εσωτερικό της Πορτογαλίας μπορεί να αποδοθούν σε μια φτωχή περιφέρεια. Γι' αυτό ε, πάντα υπάρχει ένας συσχετισμός και μια σχετικοποίηση σε σχέση με την ε, περιφερειακή συνοχή. Θεωρώ ότι οι επενδύσεις πρέπει να είναι διαφανείς, να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία και φυσικά να είμαστε υπόλογοι για τις ε, πράξεις μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθηθούν και οι πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες. Θεωρώ ότι αυτή η συμβουλευτική πλατφόρμα που προβάλλεται σχετίζεται με συνεργασία περιφερειακών τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αναδιάρθρωση αυτών των προγραμμάτων. Αν δούμε το ΑΕΠ διαφέρει πάρα πολύ ανάλογα με τις επενδύσεις σε απόλυτους αριθμούς. Υπάρχει φυσικά και μια γεωγραφική συγκέντρωση σε ορισμένα σημεία και γι' αυτό θα πρέπει όλες οι περιφέρειες ε, να έχουν ε, αυτή την προσβασιμότητα στα ταμεία με βάση αυτή τη συμβουλευτική πλατφόρμα που προβάλλουν χωρίς να υποκαταστήσει την πολιτική συνοχής. Πολλές φορές υπάρχουν ελλείψεις στην επενδυτική μας πολιτική. Θα πρέπει να πληρωθούν οι ελλείψεις της αγοράς και ο κανονισμός θα πρέπει να επεκταθεί μέχρι το 2020 για να γίνει σωστή ανάγνωση του κανονισμού και να κατανοήσουμε και το πνεύμα αυτού του κανονισμού που θα μας διέπει. Ευχαριστούμε Ζωζέ Μανουέλ. Χαίρομαι γιατί μίλησες για τις πλατφόρμες και τόνισες αυτή την τυχή του θέματος. Πολλές φορές διατάξεις που έχουμε στη διάθεσή μας δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν χρησιμοποιούνται. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ουδετερότητα ως προς την πρόσβαση. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, όπως θα καταδείξει και αυτή η συζήτηση για να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά. Ο κύριος Κάρλος Σέκη ε, είναι ο πρώτος ομιλητής από την Τέντη, είναι συντονιστής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, κυρίες και κύριοι, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Ε, πρώτον, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επίσης και διότι παλαιότερα ήμουν αντιπρόεδρος ε, της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά κάποιον τρόπο ε, επανέρχομαι λοιπόν και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η δική μου ομιλία που τη βλέπετε στη διαφάνεια σας την έχω στείλει κιόλας. Ε, θα προχωρήσω αρκετά γρήγορα θα προσπαθήσω να εστιάσω σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Πρώτα απ' όλα, έχετε μία παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα το ΕΦΣΥ γιατί αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στην περασμένη χρονιά και κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Εγώ, επειδή ακριβώ ασχολούμαι με τα προγράμματα, τα TNT, θα αναφερθώ στις ε, μεταφορές κυρίως. Και βλέπετε λοιπόν ότι οι μεταφορές, ε, παρότι είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας και παρότι εκεί είναι απαραίτητο να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις για να καλυφθούν να ε, κυρίως ε, αυτά που αφορούν περισσότερες χώρες, μιλάμε για το 10% των εγκεκριμένων κονδυλίων του ΕΦΣΙ, δηλαδή 3,6 δις και αυτό αντιστοιχεί στο 13% των ε, επενδύσεων ε, που έχουν κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ με μια μόχλευση που είναι όμως ε, αρκετά περιορισμένη ακριβώς λόγω της φύσης των προγραμμάτων για τα οποία συζητάμε. Σήμερα λοιπόν τα προγράμματα στον τομέα των μεταφορών αφορούν λιμάνια. Έχουμε το Ταμείο της Προσπελασιμότητας των Λιμανιών, όπως στην Ισπανία, ε, οδικό ε, δίκτυο σε πολλές χώρες. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ μιλάμε για το εύκολο κομμάτι ε, του ΕΦΣΥ το τροχαίο υλικό, ε, ως παράδειγμα, εδώ μπορούμε να πάρουμε την Ιταλία, να έχουμε ε, πιο ε, καθαρά αστικά προγράμματα, πράσινα προγράμματα στον τομέα της ναυτιλίας και τέλος ε, θέματα υποδομών και μετοχικό κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Για μας λοιπόν το ΕΦΣΙ πρέπει να εφαρμόζεται συμπληρωματικά στο εργαλείο Connecting Europe. Και βλέπετε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια τα στοιχεία όπου μπορούμε να δούμε τη σύγκριση ανάμεσα στο τι έχει γίνει στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ στον τομέα των μεταφορών αφενός και στις προσπάθειες ε, αφετέρου στο πλαίσιο του ΣΕΦ. Έχουμε 29 προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί. Όπως σας είπα, 2,9 εκατομμύρια. Ε, μιλάμε για τους σιδηροδρόμους, ε, για τις, ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία, το δικό δίκτυο και το ε, θαλάσσιο δίκτυο. Τώρα, το, το μέσο ΣΕΦ που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή συνδέοντας την Ευρώπη, αφορά στα κονδύλια ε, στα οποία έχουν διατεθεί. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την επιτάχυνση και μέσα από αυτήν να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες για 158 ε, προγράμματα που έχουν εγκριθεί, περίπου 45 δις είναι οι επενδύσεις και ε, το modal split είναι πολύ υψηλή ε, σημασίας ε, για τους ε, σιδηροδρόμους και Αναφέρομαι σε αυτά που είπα και προηγουμένω. Είδατε τι, τα ποσοστά στην εσωτερική πλοία και αλλού. Βλέπουμε ότι εδώ το επίπεδο είναι σκόπιμα χαμηλό, γιατί τη χρηματοδότηση μπορεί κανείς να την και αλλού. 6% οι ε, πολυτροπικές μεταφορές 43%. Και μετά έχουμε και με μονομενα προγράμματα, εκτός από τους τομείς, εκεί βλέπουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Με το ΕΨΙ το βλέπουμε αριστερά τα στοιχεία και το ε, μέσω συνδέοντας την Ευρώπη δεξιά. Στο ΕΦΣΥ προβλέπεται η στήριξη των αστικών μεταφορών. Εδώ έχουμε ε, πολύ σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν. Έχουμε τις επενδυτικές πλατφόρμες. Αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως και είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω του γεγονότος ότι έρχομαστε με το μέγεθος των προγραμμάτων και εδώ δεν υπάρχει συνέπεια με το διοικητικό κόστος που προκύπτει στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία χειρίζεται θέματα εφαρμογής. Άρα δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθούν προγράμματα και αυτό μπορεί να γίνει είτε εκ των άνω προς τα κάτω ή αντίστροφα. Στην περίπτωση που επιλέγουμε την προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω η πλατφόρμα ε, πράσινης ναυτιλίας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί εδώ μιλάμε για στάνταρτ προγράμματα τα οποία ε, μπορούν να ξεπεράσουν το διοικητικό κόστος, να μην παίζει δηλαδή τόσο μεγάλο ρόλο το διοικητικό κόστος. Μετά, την προσπελασιμότητα των λιμένων στην Ισπανία, Πόρτο, Ντελεστάντο, Consortium. Ε, εκεί λοιπόν ε, μιλάμε για ένα φορέα οποίος ε, εξετάζει το ΕΦΣΥ έτσι ώστε για να συγκεντρωθούν κονδύλια και μετά αυτά να επιμεριστούν ε, σε διάφορα μέρη για να υπάρχει ελκυστικότητα. Το pooling, το να συγκεντρώσουμε λοιπόν προγράμματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η γεωγραφική ισορροπία ε, και αυτή θα παίξει ρόλο κυρίως όσον αφορά τις χώρες συνοχής. Η μόχλευση είναι αρκετά υψηλή και στην περίπτωση του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη έχουμε μεγάλη συγκέντρωση σε ε, δύο συνοριακά προγράμματα. Έχουμε επίσης και κονδύλια τα οποία έχουν διοχετευτεί σε μικρά προγράμματα με στόχο να υπάρχει καλύτερη γεωγραφική ισορροπία παρότι έχουμε μικρότερους πολλαπλασιαστές από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις, γιατί κατ' ουσίαν μιλάμε για επιδοτήσεις ε, οι οποίες εντάσσονται μέσα και σε άλλες μορφές ε, χρηματοδότησης. Αυτό ε, που θέλω να σας επισημάνω είναι γενικότερα η προσέγγιση μας. Είπαμε ότι υπάρχει ουσιαστική συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα προγράμματα Εύση και το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν προτείνουμε όχι μία νέα, αλλά μία επιπρόσθετη προσέγγιση που την αποκαλούμε σύμμιξη. Και ε, αυτό, αν θέλετε, είναι το αποτέλεσμα και μιας, ενός διαγωνισμού, ο οποίος ε, δημοσιεύτηκε σήμερα, με στόχο να στηρίξουμε την ιδιωτική χρηματοδότηση που μπορεί να μην αρκεί και ως εκ τούτου να ε, τα συμπληρώσουμε, να συμπληρώσουμε την ειδική χρηματοδότηση με ε, προγράμματα του ΣΕΤ. Ε, έχει διαιτεθεί ένα δις και μπορεί να υπάρξει συνδυασμός με ενισχύσεις του προγράμματος ΣΕΦ ή με κονδύλια των Εθνικών Τραπεζών Δανειοδότησης ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή κονδύλια από το Έχουμε λοιπόν πολλά, ε, πολλές μορφές χρηματοδότησης και πολλών μορφών κονδύλια που μπορούν να συνδυαστούν για να βρεθεί μια λύση και για να υπάρχει ένα αποτελεσματικό χρηματοδοτικό πακέτο το οποίο κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει να εγκρίνεται πριν ένα πρόγραμμα προχωρήσει σε μια ε, διαδικασία η οποία προβλέπεται στο διαγωνισμό. Το ΕΦΣΥ θα πρέπει να χρησιμοποιείται προφανώς για να μεγιστοποιείται η μόχλευση της συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Όπως σας είπα, όλες αυτές οι λεπτομέρειες ε, μπορείτε να τις δείτε γιατί σήμερα δημοσιεύτηκαν καταληκτικές ημερομηνίε 14 ε, Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου. Πιστεύουμε, για να ολοκληρώσω και κύριο Πρόεδρε, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική δοκιμή. Είναι σαν να έχουμε ένα εργαστήριο, δηλαδή κάτι καινούριο, το οποίο υποτίθεται θα συμπληρώσει τα προγράμματα ΕΦΣΙ και ΣΕΦ και ε, είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μας ότι ε, θα πρέπει να αποκτήσουμε μέσα από αυτό το διαγωνισμό εμπειρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε και κατά την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Σέκη. Θα θερμοπαρακαλούσα τους υπόλοιπους καλεσμένους μας να μην υπερβούν το δεκάλεπτο στις παρεμβάσεις τους και να δώσω το, λόγο στον κύριο Ζουζέ Φερνάντο Φιγκερέιντορ, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του, του Χρηματοδοτικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχουμε μια πολύ σύντομη παρουσίαση για να σας δώσω κάποιες αδρές γραμμές ε, της ε, δικής μας προσέγγισης που είναι το παράθυρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα σας πω πώς το ε, προσεγγίζουμε εμείς και από την πλευρά των τραπεζών αλλά και από την πλευρά φορέων που χρηματοδοτούσαν εδώ και χρόνια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία δύο-τρεις διαφάνειες για να σας πω γιατί συστήσαμε αυτό το Ινστιτούτο Πρόθεση ε, στην Πορτογαλία που είναι ένα νεοσύστατο σχέδιο και το κάναμε γιατί ε, και στην Πορτογαλία όπως και στην Ευρώπη έχουμε ε, μια οικονομία που εδράζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ένα συντριπτικό ποσοστό της οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ψηλό τζίρο όλες μαζί και δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης. Το πρόβλημα ε, σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, γιατί ε, δεν είναι μόνο ε, πρόβλημα των χωρών του Νότου, αλλά είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, πιο οξύ βέβαια σε ορισμένε χώρε από τις άλλες Και αυτό είναι μια στατιστική παρατήρηση. Δεν είναι ποιοτική αξιολόγηση. Οι περισσότερες χώρες έχουν και πρόβλημα μετοχικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου και πρόβλημα, έλλειμμα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Και αυτό τους δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα και έλλειψη οικονομικών ροών, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες οικονομικά επιχειρήσεις και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Αυτά τα δύο προβλήματα ταλανίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το χρησιμοποιώ αυτό γιατί στη δική μας περίπτωση έχουμε το πρόβλημα ότι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμη και μεσαίες, αλλά κυρίως οι πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις, τα περισσότερα τους κονδύλια, αντί να τα επικεντρώνουν σε επενδύσεις ε, και σε αναζήτηση καινοτομίας, ε, τα αφιερώνουν στην αποπληρωμή των χρεών τους και των υψηλών επιτοκίων που χρειάζεται να καταβάλουν. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία που συγκρίνουν την Πορτογαλία με άλλες χώρες. Κατά μέσο όρο, εμείς ε, το μετοχικό κεφάλαιο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι περίπου το ίδιο σε ποσοστιαίες μονάδες με αυτό της άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε στην Πορτογαλία είναι ότι τα επιτόκια είναι πιο υψηλά. Οι τόκοι που πληρώνουμε είναι πολύ πιο υψηλοί κατά μέσο όρο από άλλους ε, Ευρωπαίους. Οπότε για μας αυτό είναι πρόβλημα, υψηλή τόκη. Βέβαια δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει τέτοιο πρόβλημα, σίγουρα και άλλες χώρες το έχουν. Γι' αυτό και αποφασίσαμε πριν από λίγα χρόνια να συστήσουμε αυτό το Ινστιτούτο πρόθεση Χρηματοδότησης ε, και αυτό ήταν ο γενεσιουργό μα λόγο. Επίση, ε, επικεντρωνόμαστε όχι μόνο σε θέματα χρέου, γιατί ο μακροπρόθεσμο δανεισμό ε, το μακροπρόθεσμο χρέο είναι πρόβλημα, αλλά και η κεφαλαιοποίηση είναι πρόβλημα, ή το μετοχικό κεφάλαιο, ή το ιονή μετοχικό κεφάλαιο στην αναζήτηση των χρηματοδοτικών λύσεων. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμαστε και με άλλους χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες που είναι είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι, δημόσιοι φορείς. Συνεργαζόμαστε με τράπεζες, εγκυτικά ταμεία και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε μια χαρτογράφηση του στρατηγικού μας σχεδίου και όπως βλέπετε έχουμε και τις δραστηριότητες μας με διαχείριση διαρθρωτικών κυρίως κονδυλίων και τις ε, μη κοινοποιημένε δραστηριότητες για τα υπόλοιπα κονδύλια. Και εδώ, όπως και στο προηγούμενο παράθυρο, έχουμε δυνατότητα χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ και όπως είπαν και οι συγκητές, θα ήταν καλό στην επόμενη φάση είναι ακριβώς να προωθήσουμε στις χώρες που είναι χώρες συνοχής, στις περιφέρειες που είναι περιφέρειες συνοχής, να προωθήσουμε τη δυνατότητα συνδυασμού των διαφόρων χρηματοδοτικών πηγών για να έχουμε μόχλευση στα χρήματα των φορολογουμένων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και βλέπετε στη διαφάνεια τα επιμέρους σημεία. Έχουμε και ε, κοινοποιημένα και μη κοινοποιημένα, γνωστοποιημένα και μη γνωστοποιημένα παράθυρα. Επίσης εδώ έχουμε τον τρόπο διαχείρισης και της, ε, το, δαν, δανεισμό. Έχουμε ε, τα 500 εκατομμύρια ε, το μέσο του ΕΦΣΥ ή το, του ορίζοντα 2020 και να περάσω τάχη στα συμπεράσματα και στις συστάσεις. Δύο πολύ σύντομε διαφάνειες από την πείρα και τις παρατηρήσεις μας έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα χρησιμοποιώντας και την πείρα και άλλων ε, παρόμοιων φορέων. Θεωρούμε ότι ε, το μέλλον του ΕΦΣΙ έχει να αντιμετωπίσει κάποιες προκλήσεις. Και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ για να διευρύνει τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου. Η πρώτη πρόκληση είναι να έχουμε αρκετή δύναμη πυρός, δηλαδή αρκετά χρήματα που να καλύπτουν τη ζήτηση. Και σε ό,τι αφορά το παράθυρο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, ζήτηση υπάρχει. Δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσει και οι μεσαίε επιχειρήσει ε, χρειάζονται χρηματοδότηση, ψάχνουν κονδύλια ε, που φυσικά θα συνάδουν με του στρατηγικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώ δεν θα, θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό και χαιρετίζω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, από πέρυσι το Σεπτέμβριο για αύξηση του προπολογισμού. Οι προκλήσεις πάντως είναι υπαρκτές. Χρειάζονται ε, επαρκή πόροι για να προχωρήσει το Ταμείο. Πέραν όμως αυτής της πρώτης πρόκλησης, υπάρχει κάτι άλλο που αναφέρθηκε. Η δεύτερη πρόκληση, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα δίκτυα θεσμικών οργάνων και φορέων που δραστηριοποιούνται επί τόπου και γνωρίζουν καλά την κατάσταση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γνωρίζουν το νηστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γνωρίζουν τι κάνουν οι επιχειρηματίε, γνωρίζουν τι συμβαίνει και θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξετάσουμε αυτό το δίκτυο θεσμικών φορέων που υπάρχουν και να το χρησιμοποιήσουμε, να το αξιοποιήσουμε αντί να δημιουργήσουμε νέα ταμεία που λαμβάνουν υπόψη μάκρο υποδομές και δεν γνωρίζουν την κατάσταση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. γιατί μερικές φορές ε, δρομολογούνται τα κονδύλια μέσω των πιο αποτελεσματικών εντό εισαγωγικών τραπεζών, αλλά αυτό δεν είναι πάντα ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν ε, οι αδυναμίες της αγοράς. Μία άλλη πρόκληση που ήδη επισημάθηκε αφορά την προσθετικότητα και την ε, καταμέτρησή της, την αξιολόγησή της ε, στη χρήση των κονδυλίων. Και μάλιστα σε μια επιτροπή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χρηματοδότηση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ακριβώς κάνουμε αυτό που και εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια φόρμουλα για να ποσοτικοποιούμε την προσθετικότητα. Αυτό είναι πρόβλημα παντού στον κόσμο. Θέλουμε, αναζητούμε έναν τρόπο για να δούμε πώς θα ορίσουμε επιτέλους την προσθετικότητα και να την αποδεχτούμε και να μπορούμε να την καταμετρήσουμε κιόλα. Γιατί οι τράπεζες ή άλλα εγγυητικά ιδρύματα χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια για να έχουν νέες πηγές χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεσαίες, τα mid-caps. Ε, και το κάνουν αυτό όντως ε, και συμβάλλουν αυτά τα κονδύλια για να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της αγοράς ή όχι. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και πρόκληση. Επίσης, μια, ένα άλλο ζήτημα συναφές με το προηγούμενο, υπάρχει ανάγκη ενίσχυση του συντανισμού ε, μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων. Ε, γιατί καλό είναι να γίνεται η σωστή διανομή, αλλά να εξασφαλίζεται σωστό συντονισμό και με του τοπικού και περιφερειακού εταίρους ώστε να έχουμε μια πραγματική κάλυψη εδαφική στις ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες και να φροντίσουμε ώστε τα κονδύλια αυτά που είναι ουσιαστικά κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογουμένων να φτάνουν σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις περιφέρειες που υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν επιλέξιμα προγράμματα, επιλέξιμα με βάση τους στόχους της Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι σκόπιμο και από άποψη πολιτικής. Επίσης, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία αυτό που ήδη υπάρχει σε χρηματοδοτικά μέσα και μέσα πρόθεσης. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό ε, και να επινοήσουμε νέες λύσεις. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε ήδη θετικές λύσεις που έχουν αποφέρει καρπούς στο παρελθόν. Και επίσης να δημιουργήσουμε μικρούς πόλους και αυτούς να αξιοποιήσουμε, όπως συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο πολλές φορές. Αυτές είναι οι προκλήσεις, απλούστευση, χρησιμοποίηση των ήδη εφισταμένων δομών και αξιοποίησή τους και επίσης ως προς τις προκλήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό εξετάζουμε τώρα. Και στην περίπτωσή μου, στο παράθυρο δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δεύτερη πρόκληση είναι, και αυτή είναι και η σύστασή μου, να δοθεί σαφής προτεραιότητα στη χρήση των, στην αξιοποίηση των ε, εφισταμένων δομών ε, του μετοχικού κεφαλαίου, των εταιρικών σχέσεων, των τραπεζών, των ε, διαφόρων χρηματοπιστωτικών δομών δικτύων όπως ε, ο κόμβος αυτός παροχής επενδυτικών συμβουλών, ώστε να ενισχυθεί και η ζήτηση ταυτόχρονα. Και αυτό ε, συνδέεται με το τρίτο εδάφιο. Σίγουρα χρειαζόμαστε υψηλή μόχλευση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η μόχλευση σημαντική. Γιατί ε, μιλάμε για 20 πλάσια, 30 πλάσια, 30 πλάσια μόχλευση. Ναι, μεν, χρήσιμο αυτό, αλλά δεν αν δεν έχουμε και τα ποιοτικά αποτελέσματα του πολλαπλασιαστή, αν ε, έχουμε με μια εγγύηση 2% τότε θα έχουμε πολλαπλασιαστή ε, πολύ μεγαλύτερο. Αλλά αυτό δεν είναι κατά ανάγκη η απόδειξη ότι αξιοποιούμε σωστά τα κονδύλια. Θα πρέπει αυτό πρώτα να κοιτάξουμε ποιοτικά ε, ποια είναι η επίπτωση και η προσθετικότητα είναι απαραίτητη και η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ποιοτική πτυχή και τη, τους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το σχεδιασμό των διαφόρων μέσων. Και ένα από τα πράγματα που παρατηρούμε στο δικό μας έργο είναι ότι μερικές φορές έχουμε κάποια προϊόντα που ε, δίνονται σε μακροεπίπεδο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά όταν φτάνουμε σε τοπικό επίπεδο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις κρατικές ενισχύσεις. Και οι μηχανισμοί του Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Ταμείων ή της ΕΤΕ δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Προσοχή όμως, προσοχή σε αυτό, γιατί μερικές φορές ε, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα παρόλο που έχουμε τη δυνατότητα μερικές φορές. Προσκρούμε σε, άλλους, ε, σε άλλα εμπόδια. Απλά λοιπόν, απλά και συνδυασμό στο μέτρο του δυνατού με τις υπόλοιπες ε, χρηματοδοτικές δυνατότητες και τα υπόλοιπα μέσα. Βεβαίως θα ε, αποζητήσουμε μία φόρμουλα για την προσθετικότητα, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Ο κύριος Μπέρναρτ Ζαγκμάιστερ που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκυοδοσίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αξιότιμε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά γιατί φέτος η δική μας η Ένωση, η ΑΤΣΕΜ, ζει και ορτάζει τα 25 χρόνια της. Αυτά τα 25 χρόνια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με τους διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε λοιπόν μέλη τα οποία είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως και άλλους που δεν είναι μη κερδοσκοπική, άρα δηλαδή μπορούν να είναι κρατικοί ή μη κρατικοί ή και αμυγός ιδιωτικοί φορείς. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλοι μας οι φορείς ε, με τα προγράμματα εγκυοδοσίας ε, επιδιώκουν τους ίδιους στόχους όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή καινοτομία, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Τώρα, με το ΕΦΣΥ Μέχρι πέρυσι υπολογίσαμε ότι με τα μέλη μας έχουμε συμβάλει κατά 25% στην επιδίωξη των στόχων. Δηλαδή το 84% των επενδύσεων ε, έχει δικινητοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Μιλάμε για 69 εκατομμύρια ε, στηρίζονται 400 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 25% εξ αυτών είναι πελάτες των δικών μας των μελών. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση την τελευταία δεκαετία. Ε, έχουν αυξηθεί οι εξασφαλίσεις που ζητούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Άρα δηλαδή ε, μιλάμε για μια μεγάλη πρόκληση. Παρόλα αυτά όμως ε, το να αποφεύγονται οι κίνδυνοι με τη ρύθμιση των ε, τραπεζών αυτό πράγματι ε, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τις, ε, τη ρύθμιση των τραπεζών υπάρχει και το περίφημο funding ratio που τι σημαίνει, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάθε φορά μόνο και μικρότερη διάρκεια, άρα δηλαδή αυτό συνεπάγεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως όταν εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα, ε, χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους. Αυτό είναι μια μεγαλύτερη δυσκολία. Εδώ προστείται και το θέμα των επιτοκίων. Τα επιτόκια είναι χαμηλά, οι τράπεζες υφίστανται πίεση Άρα δηλαδή κυρίως σε μικρά προγράμματα οι τράπεζες, ε, για τις τράπεζες δεν είναι πλέον δυνατό ε, να επιτύχουν μεγάλα κέρδη ως εκ τούτου αυτά τα μικρό προγράμματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν σχέση με νεοφυρείς επιχειρήσεις ε, είναι δύσκολα αυτά να χρηματοδοτηθούν άρα δηλαδή χρειαζόμαστε εδώ κονδύλια. Όπως και για τους προαλήσεντες για μας πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντα συνδυασμό με το πρόγραμμα ΕΨΗ. Και εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω ε, ιδιαίτερα τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, κυρίως με το EIF, ε, με τα δύο προγράμματα Κόσμο και Inofin. Αυτά τα δύο προγράμματα είναι σημαντικά για μας. 16 μέλη μας από 13 χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ για αυτά τα εργαλεία εγκυοδοσίας. Όμως θέλω να σας πω ότι έχουμε και πολύ μακρά εμπειρία. Πριν από το ΕΦΣΥ Είχαν και άλλα πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, χαρήκαμε ιδιαίτερα που τον Ιούλιο του 2016 ε, χρησιμοποιήθηκαν 500 εκατομμύρια από τις καινοτομίες μετακινήθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς επιθυμούμε τώρα πλέον να διεκδικήσουμε το διπλασιασμό των κονδυλίων. Ε, εξάλλου ε, κάναμε μια ε, δημοσκόπηση, ένα ερωτηματολόγιο, στείλαμε στα κράτη-μέλη, στα κράτη -μέλη, στους, στους, οργανισμούς μας και έχουμε διαπιστώσει ότι μέχρι το 2020 υπάρχει ε, ζήτηση για περίπου 3 δις ε, εγγύσεων. Αυτό πρέπει να σου πω μας απασχολεί γιατί και κατά τους επόμενους μήνες θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η νέα προσφορά θα καλύπτει και τη ζήτηση. Μιλάμε για τη ζήτηση εκείνη που αφορά τις counter guarantees αλλά όχι τις άμεσες εγγύησεις. Εμείς ως Ένωση αυτή τη στιγμή έχουμε αναθέσει μία μελέτη στην KPGM στην Ιταλία. Η μελέτη αυτή είναι έτοιμη, μας την έδωσαν και τώρα λοιπόν μπορέσαμε να κάνουμε μία σύγκριση για το ε, ποια είναι η διαφορετική επίδραση των δύο διαφορετικών διάβλων. Δηλαδή κατά πόσον οι εγγυήσει θα πρέπει να δίδονται άμεσα από τις τράπεζες ή κατά πόσον οι εγγυήσει θα πρέπει να δίνονται από φορείς εγκυοδοσίας, εθνικούς και περιφερειακούς. Υπάρχουν αυτές οι δύο διαφορετικές δυνατότητες εγκυοδοσίας. Και ε, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία συζητήσαμε, ε, τα συζήτησαν τα μέλη μας και διαπιστώσαμε ότι οι counter guarantees ε, πειράζουν πολύ περισσότερο την απασχόληση και την καινοτομία, πολύ περισσότερο από ότι οι εθνικές και οι περιφερειακές εγγύσεις. Οι εμπορικές ε, τράπεζες εστιάζουν κυρίως σε εμπορικά προγράμματα. Όταν πρόκειται για μακροοικονομικά προγράμματα, οι ε, άλλες εγγύησεις είναι πολύ πιο σημαντικές. Αυτό που ενδιαφέρει είναι και τα ενωσιακά κονδύλια, γιατί αυτά εμπλουτίζονται και με εθνικά κονδύλια και με τον τρόπο αυτό προκύπτει μια μεγαλύτερη μόχλευση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγων είναι ότι η ε, εγκυοδοσία αφορά όλες τις τράπεζες και όχι μόνο λίγες όπως συμβαίνει με τις ε, άμεσες εγγύσεις. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν, δεν προκύπτει στρέβλωση της αγοράς. Ε, κατά την άποψή μας και λόγω του ότι υπάρχουν αυτά τα πλεονεκτήματα σε ε, μακροοικονομικά προγράμματα ε, θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε τις counter guarantees και να τις προτιμούμε από τις ε, άμεσες εγγύησεις γιατί αυτές έχουν πολύ καλύτερη μόχλευση. Συγκεκριμένα μέτρα είναι στις περιπτώσεις όπου οι εγγύησεις συνοδεύονται με τέλη όπως το Inofin θα πρέπει να ε, έχουμε κατά νου την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δωρεάν, όπως το πρόγραμμα COSME, τότε όταν επιλέγονται οι ενδιάμεσοι θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε counter guarantees, σε εθνικούς ε, και περιφερειακούς ε, φορείς ε, εγκυοδοσίας, γιατί ακριβώς προκύπτει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Για το COSME προτείνουμε 150 ευρώ ως κατώτατο όριο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε καινοτόμα και σε μη καινοτόμα προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κατώτατο όριο, γιατί θεωρούμε ότι με αυτό θα διευκολυνθεί κατά πολύ η εφαρμογή των προγραμμάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να υπάρχει υποχρέωση ε, λογοδοσίας, ε, διαφάνεια και όπως και οι προλαλήσαντες και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά τις άμεσες εγγυήσει και τις counter guarantees δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση και καμία διακριτική μεταχείριση ανάμεσα στις δύο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το πρόγραμμα FC2 ε, προγραμματίζεται διότι το πρόγραμμα των, των εγγυήσεων ε, ε, προκαλεί μεγάλη μόχλευση και να επισημάνω επίσης ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους ενδιάμεσους λειτουργεί θαυμάσια και γι' αυτό επιτρέψτε μου με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστώ θερμά όλους αυτούς τους θεσμούς. Θέλω όμως να επισημάνω ότι αυτή η σημαντική μόχλευση δεν αρκεί, διότι η μόχλευση δεν έχει πάντα άμεση σχέση με μακροοικονομικές επιπτώσεις, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενδιάμεσοι φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζαμάρα Ρουζουτζίντλο έχει το λόγο, ε, η οποία είναι Διευθύνων Σύμβουλο στο Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνεισηγητές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι γιατί μπορώ να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μας ε, μέσα στα πλαίσια του ΕΦΣΥ Θα ήθελα να σταθώ ε, στην πλευρά του προγράμματος και του φορέα προώθησης και τη συνδεσιμότητα σε σχέση με τη χρηματοδότηση του ε, δημόσιου τομέα ως προς ε, εμπορικές επιχειρήσεις. Φυσικά υπάρχει οπωσδήποτε θετική ανταπόκριση από τους ε, ενδιάμεσους, από τους μεσάζοντες ε, σε σχέση με την διαδικασία σύμβασης διάθεσης των προϊόντων προς την αγορά και υπάρχει μία ευελιξία για να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Ε, Επίσης υπάρχει μία ορατότητα ως προς τα στοιχεία που θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και και φυσικά αυτό το μέσον μπορεί να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και καινοτόμα στοιχεία ορισμένων προγραμμάτων, άρα θα κινηθούν πέρα από το προγραμματισμένο χρονικό πλαίσιο γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν μακροχρόνια. Και φυσικά χρειάζεται περαιτέρω απλούστευση ε, ως προς τις ε, κοινέ προσπάθειες και συνδεσιμότητα του ΕΦΣΙ με το, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει απόλυτη ανταπόκριση από τα προγράμματα και υπάρχουν και επιπρόσθετα προγράμματα και γι' αυτό αυτή, αυτό το στοιχείο προσθετικότητας δεν χρηματοδοτείται. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ε, διαφάνεια για τις τροποποιήσεις που θα επέλθουν. Γιατί πολλές φορές λαμβάνω πληροφορίες για κάποια αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά δεν υπάρχουν ε, σημεία διείσδυσης των ίδιων των φορέων σε σχέση με τις ε, λύσεις που μπορούν να προβληθούν και περαιτέρω πληροφορίες οι ε, στόχοι διάδοσης στα κράτη-μέλη υπάρχουν και καταλαβαίνετε ότι εκπρόσωποι από τα Υπουργεία προσπαθούν να διαβλέψουν την όλη διαδικασία έτσι ώστε να φτάσουμε ε, στην συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού φορέα, αλλά πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία. Ως προς τις ε, περαιτέρω εξελίξεις, αυτό που έχει σημασία είναι η προσθετικότητα ε, του ΕΦΣΥ με της ΜΜΕ, αυτού του διάβλου. Ο προσθετικός χαρακτήρας είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να βρούμε και έναν ορισμό για την προσθετικότητα. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος ε, ορισμός. Θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσο αυτή η διάβλη με τις ΜΜΕ είναι αρκετά ευέλικτη. Για να δούμε κατά πόσο και το έτσι μπορεί να προβάλλει μία συγκεκριμένη χρηματοδότηση με μειωμένη γραφειοκρατία. Αν δούμε όμως τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, εδώ υπάρχουν ε, λειτουργικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία σχετίζονται και με χρηματοδοτικά ε, μέσα στα πλαίσια των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Στο σχέδιο Juncker έχουμε όριμους καρπούς, από όσο φαίνεται, και τη στιγμή που θα αρχίσει να δρά το εύση θα είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστούμε τα χαρτοφυλάκια και το 2018 θα ρωτηθούμε πώς ε, δαπανίσαμε τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια του crowding out και αυτό που έχει σημασία είναι και η σύμιξη των ε, ταμείων και πώς μπορούν να δράσουν στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνία μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Να δούμε δηλαδή τις πρακτικές που προϋπάρχουν στην αγορά μέσω ΕΤΕ, υπομνημάτων ΕΤΕ, σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ανάλυσης κόστους ωφελίας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι προϋπάρχει στην αγορά για να γίνει χρηματοδότηση μέσω του σχεδίου Juncker και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν ελλείψεις θα πρέπει να υπάρξουν κατά, περίπτωση, προγράμματα για να ενισχυθούν και άκουσα από πολλούς φορείς ότι δεν ήξεραν ότι έχουν πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών γιατί δεν ήξεραν το σχέδιο είναι έτοιμο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο στην ιστοσελίδα υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες. Αν λοιπόν ο επικεφαλής του σχεδίου μιλήσει με τον υπεύθυνο ενός ε, διαρθρωτικού επενδυτικού ταμείου και κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη δυνατότητα αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι επιτόπια τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των στοιχείων, των επενδυτικών στοιχείων και της επιλεξιμότητάς τους δυνάμει του εύση και των ΕΔΕΠ, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Πολλές φορές οι επικεφαλής των σχεδίων έκριναν, μάλλον τους ελέγχθη ότι θα έπρεπε να υποβάλουν δύο αιτήσει δυνάμει του σχεδίου Juncker και, τις, και επιμέρους χρηματοδοτήσεων, διότι υπάρχουν θέματα επιλεξιμότητας. Αν λοιπόν μιλάμε για προσθετικότητα ως προς την ε, χρηματοεπενδυτική δραστηριότητα θα πρέπει να προβάλλουμε σχέδια χαμηλότερου κινδύνου, διότι μιλάμε για μία άλλη ροή χρημάτων με μία διαφορετική προετοιμασία. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιλογές blending αυτής της διαδικασίας σύνηξης, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές επιδοτήσεις, την ε, διαχείριση των χαρτοφυλακίων, τις συμβατικές λύσεις και ούτω καθεξής. Ήδη έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για αυτό το blending του ΕΦΣΙ και των ΕΔΕΠ e αν δείτε όμως αυτό το έγγραφο, δεν έχετε σαφείς πληροφορίες. Με βάση λοιπόν αυτά τα σχέδια και με τις ε, επιμέρους μετατροπές βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν οι προσμίξεις που πρέπει με βάση τα χρηματοεπενδυτικά σχέδια πρέπει να προβάλλουμε μία βαθύτερη διαδικασία. Ξέρω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί ε, δεν διέπονται από ευελιξία, αλλά αν δεν ξεπεράσουμε αυτή την στενοπό, τότε μόνο οι συμβουλευτικές εταιρείες θα μας βοηθήσουν. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής προγραμμάτων από την ΕΤΕ. Θυμάμαι το Μάρτιο πέρσι συζητήσαμε το ίδιο θέμα και δεν έχει επιτελεστεί καμία πρόοδος από τότε. Άκουσα και για περιπτώσεις όπου το σχέδιο Juncker για επιμέρους προγράμματα προβάλλει τον ίδιο τύπο χρηματοδότησης με την ΕΤΕ. Απλώς υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Από όσο κατανοώ δεν ήταν αυτός ο στόχος μας. θέλουμε να προωθήσουμε καλύτερα τη χρηματοδότηση, να υπάρχουν επιμέρους εγγυήσεις και καλύτερες εγγυήσεις, αλλά αν θέλουμε να είμαστε πιο καινοτόμοι και να μην κινούμαστε με βάση το διαρθρωτικό χαρακτήρα, θα πρέπει να υπάρχουν επιλογές επιμερισμένου κινδύνου. Αν δούμε τις δυνατότητες της ΕΤΕ, πολλές φορές υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου. Άρα ίσως το, αυτή η επιχειρησιακή αποτίμηση δεν είναι σωστή. Ίσως θα πρέπει να γίνεται μια διαφορετική αξιολόγηση με βάση το σχέδιο Juncker. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες της ΕΤΕ. Επίσης θα πρέπει να ε, εξευρεθούν καλύτερες λύσεις επιμερισμού του κινδύνου με βάση τον προσθετικό χαρακτήρα του ΕΦΣΙ. Ακριβώς αυτό είπα και προηγουμένως, στο προηγούμενο σημείο δηλαδή. Δηλαδή αυτό που μας ενδιέφερε ήταν στην ΕΤΕ να έχουμε συγκεκριμένες επιλογές επιμερισμού κινδύνου που να αναλαμβάνουν οι μεσάζοντες. Καλύτερη επικοινωνία επίσης για την διαδικασία επιλογής των σχεδίων. Πρέπει να τελειώσω. Ναι, σας παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσετε. Ε, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα ήταν απόλυτα σαφές και είναι τροφή για συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ ε, χρήσιμα αυτά που μας είπατε και μας εμπνέουν και τροφοδοτούν την περαιτέρω συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Χαργιτάη που είναι διευθύντρια στο τμήμα Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Συγχρηματοδότησης και Χρηματοοικονομικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε που έχω την ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας γιατί η τράπεζά μας, η ΕΤΑ, είναι η τράπεζά σας που ανήκει κατά κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και στην ΕΤΕ. Ε, ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια για να πραγματοποιήσει ε, επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Είμαστε παρούς, παρόντες σε 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είμαστε στο ΕΦΣΙ, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων. Είμαστε ταυτόχρονα δηλαδή insider και outsider. Είμαστε εντός, εκτός και επιταυτά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ε, και θα ήθελα σε ένα λεπτό να σας πω που έγκυται οι διαφορές μας. Καταρχήν εμείς ε, δραστηριοποιούμαστε τοπικά. Επαναλαμβάνω, Έχουμε 110 περίπου τραπεζικούς σε 12 χώρες. Έχουμε συμβούλους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 90% των επενδύσεών μας στις χώρες αυτές που ξεκινάνε από την Ελλάδα, την Κύπρο, Λιθουανία, Εστονία. Εκεί συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις. Επίσης, ε, πολλοί αναφέρθηκαν ε, σε μεγάλα, επίβολα σχέδια. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε μικρότερα σχέδια, 20 εκατομμυρίων ε, ευρώ. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Επίσης, έχουμε από την αρχή της ίδρυσής μας ε, να αναλαμβάνουμε και κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιό μας, τον ηχοστολογιζό μας. Και μάλιστα πήραμε μετοχικό κεφάλαιο από ελληνικές τράπεζες. Φαντάζεστε πόσο, ε, τι όρεξη έχουμε για κίνδυνο στην ΕΤΑ. Επίση, προσθετικότητα. Προσθετικότητα σε σχέση με τι ε, επενδύσει των εμπορικών τραπεζών. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια με την Unicreditor, γιατί αλλιώ ε, η, μέτοχοι θα έρθουν και θα παραπονεθούν. Εμεί θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα συγκρότηση και Ανάπτυξη. Και όταν συνεργάζομαι με του πελάτε μου, θα πρέπει να του ε, ενθαρρύνω, να του σωθώ. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, να βρουν γυναίκες, επιχειρηματίες, να κάνουν τη διαφορά. Επίσης η τράπεζά μας προσπαθεί να μεταμορφώσει το επενδυτικό περιβάλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την επιτυχία του ΕΦΣΥ να προωθήσει περαιτέρω τις ε, εταιρείες στήριξη, τις ε, προσπάθειες στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον. Αυτό κάνουμε και εμείς τουλάχιστον σε 12 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επίσης ε, προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας στις ανάγκες των πελατών. Δεν έχουμε μαζική παραγωγή, αφουγκραζόμαστε του τους πελάτες, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί τόπου, Συνεργαζόμαστε με ντόπιου συμβούλου, ε, στηρίζουμε ευρηματικέ δημιουργικέ βιομηχανίε για να ετοιμάσουν το επενδυτικό του σχεδιασμό, στηρίζουμε γυναίκε επιχειρηματίε και φυσικά και πράσινη ανάπτυξη. Πέρυσι είχαμε 33% των επενδύσεών μα που συνέβαλε σε ε, δραστηριότητες υπέρ του κλίματος ε, και ο στόχο μας είναι το 40%. Και χρησιμοποιούμε δικά μας κονδύλια, οπότε ε, το κέρδο που αποκομίζουμε το αφιερώνουμε στις δραστηριότητε μας σε 12 χώρε μέλη. Και δεν έχουμε πρόσβαση σε ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δεν επωφελούμαστε από επιχορηγήσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, από τι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί δραστηριοποιούμαστε σε 12. Και μάλιστα κάποιο συνάδελφο από την Ρουμανία με ρώτησε αν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα σχέδια και να περιλάβουμε περισσότερες ε, χώρες. Περιμένουμε περισσότερα προγράμματα από τις χώρες αυτές. Θέλουμε να προετοιμάσουμε ΣΔΙΤ, ε, σχέδια υποδομών, ε, βοήθηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτα εσείς θα πρέπει να κάνετε την προεργασία και μετά να μπει η ΕΤΑ και να βοηθήσει περαιτέρω. Επίσης, να δώσουμε το καλό παράδειγμα και σε άλλους για να μιμηθούν αυτή την εμπειρία. σε τι επικεντρωνόμαστε. Φυσικά δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα αλλά σίγουρα ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, βιώσιμη αστική κινητικότητα, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στι υποδομέ. Αυτά τα λέω επιγραμματικά. Δεν είναι εξαντλητικό ο κατάλογο. Πάντω έχουμε συγκεκριμένη επικέντρωση σε ε, είδη επενδύσεων. Ε, ε, μας αρέσει ο κίνδυνος, χρησιμοποιούμε και τις εγγύησεις, έχουμε λιγότερο από 10% ε, των, ε, της χρηματοδότησης ε, λαμβάνουμε κρατικές εγγύησεις και επίσης συνεργαζόμαστε και με τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία. Μάλιστα έχουμε τώρα 120 εκατομμύρια ευρώ δάνεια στη Βουλγαρία και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μόχλευση με την δική μας χρηματοδότηση. Αλλά έχουμε κάποιες δυσκολίες και εμπόδια που θα πρέπει να υπερκεράσουμε. Επίσης, ε, έχουμε κάποια διάρθρωση μετοχικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Λιθουανία και δίνουμε συμβουλές στι λιθουανικές αρχές για τη διαχείρισή τους, αλλά ταυτόχρονα είμαστε εντός και εκτός, οπότε περισσότερο ασχολούμαστε με τη διευθέτηση των θεσμικών σχέσεων παρά με τη συμβουλή για τη διαχείριση. Πάντως, ε, έχουμε πολλέ συχνά επαφέ με το ΕΦΣΥ. Και μάλιστα Είχαμε μια ΣΔΙΤ Σλοβακίας ε, και Λιθουανίας ε, για ένα οδικό δίκτυο και συνεργαζόμαστε με την ΕΤΕ. Το ίδιο και στην Ελλάδα για συναλλαγές υψηλού κινδύνου. Όπω σας είπα η ΕΤΑ έχει αναλάβει υψηλό κίνδυνο στην Ελλάδα με, ε, κάποιες, με κάποια εγγυημένα δανειακά ομόλογα. Επίσης επενδύουμε και σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και περιμένουμε περισσότερα ε, προγράμματα από τη Ρουμανία, Κροατία, Ελλάδα σε υποδομές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Εκεί θα χρηματοδοτήσουμε με το συνήθι εταιρικό κίνδυνο. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο όμως είναι η επόμενη διαφάνεια, γιατί πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να ε, να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά. Και Είχαμε ήδη συνεργασία με τις υπηρεσίες στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και συνεργαζόμαστε στις, χώρες του, στις 12 χώρες ε, και στα θέματα διαχείρισης των μη εξυπηρετωμένων δανείων. Ε, επίσης, θέματα ε, ένωση κεφαλαγορών. Έχουμε σχετικά προγράμματα στη Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία και Κροατία. Θέλουμε να συνεργαστούμε σε θέματα μεταρρύθμιση πολιτικών για να προωθήσουμε την ενεργειακή απόδοση, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις υποδομές, είναι επιλογή πολιτικής εδώ, και επίσης συνεργαζόμαστε με ένα σχέδιο που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε από κοινού στις χώρες αυτές, ό,τι αφορά τις επενδυτικές πλατφόρμες, και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς θα, θα, θέλαμε περισσότερες επενδυτικές πλατφόρμες, πανευρωπαϊκές. Οι χώρες ζητούν και εθνικές ε, πλατφόρμες, γιατί όταν είναι πανευρωπαϊκές πλατφόρμες ε, ε, τα έχουν κάπως χαμένα οι χώρες. Αλλά και ίσως και τοπικές και περιφερειακές πλατφόρμες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί επικεντρώνονται συγκεκριμένες χώρες και επίσης οι κίνδυνοι μπορεί να ε, μεταδοθούν στην Ευρώπη, αλλά έχουν ιδιαίτερα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά. Οπότε μας ε, θέλουν να τους παρουσιάζουμε το φάσμα κινδύνων που βρίσκεται στη, στο στόχο μας. Επίσης, μας ενδιαφέρει η ενεργειακή απόδοση και σχετικά προγράμματα. Επίση, δεν μιλώ πολύ για εθνικέ ε, τράπεζε πρόθεση, γιατί δεν, συνεργόμαστε μαζί, δεν συνεργαζόμαστε μαζί του. Συνεργαζόμαστε με τι εμπορικέ τράπεζε. Τα δικά του χρήματα θέλουμε στι πλατφόρμε. Επίση, έξυπνε πόλει μπορούν να χρηματοδοτηθούν με εμπορική βάση, με συμμετοχή του ΕΦΣΥ, με συμμετοχή τη ΕΤΑ και χρηματοδότηση από τι ε, εμπορικέ τράπεζε ε, ή εθνικά Ινστιτούτα Προώθηση. Άρα θέλουμε και χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και πολύ ευχαριστώ να προετοιμάσουμε στήριξη της προετοιμασίας των σχεδίων και χρηματοδότησή τους. Επίσης, άμεση χρηματοδότηση με τους συναδέλφους της ΟΕΤΑ. Έχουμε εταιρείε που έρχονται και ζητούν χρηματοδότηση βρυδική, τύπου μεζανίν. Ε, και εκεί προσπαθούμε να βρούμε τα κενά που υπάρχουν στι χώρε αυτέ και να τα καλύψουμε για να έχουμε καλύτερη διάρθρωση των ε, επενδύσεων στι υποδομέ. Επίση έχουμε διαπραγματεύσει και με τον κόμβο παροχή επενδυτικών ε, συμβουλών. Γιατί εμείς έχουμε τις σωστέ υπηρεσίες για παροχή επενδυτικών συμβουλών στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό το έχουμε αποδείξει η Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Εμεί έχουμε μεθοδολογία και συνεργαζόμαστε με τοπικού συμβούλου. Οπότε δεν ισχύει αυτό το με ένα σπάρο δύο τριγώνια, αλλά έχουμε μεγάλη έκταση μεν, αλλά ε, δίνουμε έμφαση στι ντόπιε επιχειρήσει, στου ντόπιου συμβούλου, γιατί αυτοί δίνουν και πιο ποιοτικέ συμβουλέ. Οπότε χρησιμοποιήστε μα. Έχουμε το εύρο στην κάλυψη και μπορούμε να ε, συμμετέχουμε στο ΕΦΣΥ με εντοπισμό και αναδιάρθρωση των σχεδίων, γιατί είμαστε παρόντες στις χώρες αυτές. Οπότε θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και με, με εταίρους που θα χρησιμοποιούν τις εγγυήσεις του ΕΦΣΥ και θα μπορούν να λαμβάνουν περισσότερους κινδύνους είτε μέσω των επενδύσεων είτε μέσω επενδυτικών πλατφορμών. Και πολύ ευχαρίστω να συμβάλλουμε στην προετοιμασία σχεδίων και προγραμμάτων υποδομών. Το κάναμε. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, ετοιμάσαμε τα πρώτα 7 προγράμματα για έξυπνες πόλεις και κινητικότητα ε, στις πόλεις, χωρίς ε, κρατικές εγγύησεις και χωρίς εγγύηση από το, από το ΕΦΣΙ. Και παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Οπότε μπορούμε αντίστοιχα αποτελέσματα να έχουμε και σε άλλες χώρες και ευχαρίστω να συνεχίσουμε να, να, ξεπεράσουμε το θέμα των, της παροχής συμβουλών μόνο στι μικρομεσαίες επιχείρησει. Επίση, μπορούμε να βελτιώσουμε τι επενδυτικέ συνθήκε στη συνεργασία με του εταίρου, γιατί έχουμε πολλέ καλέ τράπεζε στι χώρε αυτέ, μέσω τη κοινοπραξία, διαφόρων ταμείων και τη παράλληλη χρηματοδότηση, μπορούμε να τι συμπεριλάβουμε και αυτέ τι εμπορικέ τράπεζε, για να μην νιώθουν απομονωμένους. Οπότε νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη είναι πολύ καλό εταίρο στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, πέντε εμπειρογνώμονες ε, για τις επεξηγήσεις αυτές. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια προόδου για περαιτέρω πληροφόρηση, απλούστευση και φυσικά η μεγάλη ικανοποίηση είναι η απασχόληση. Χρειάζονται σύμβουλοι για ενημέρωση, για παροχή συμβουλών και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους και καταρχήν θα δώσω το λόγο στους εισηγητές, συνεισηγητές Ισκιώδης στην κοινή, στη, στη Joint Committee, την κοινή Επιτροπή Προϋπολογισμών και ε, Οικονομικών Υποθέσεων και καταρχήν θα δώσω το λόγο στον Ούτο Μπούλμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κοιτάξτε, ε, εάν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους συναδέλφους που δεν είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν, ε, θα προτιμούσα να μιλήσουν εκείνοι και εσείς αν θέλετε μπορείτε να μου ξαναδώσετε το λόγο ε, στην κατακλίδα της σημερινής συνεδρίας. Ό,τι θέλετε κύριε Πρόεδρε, αποφασίστε εσείς. Εάν επιθυμείτε, έχετε το λόγο ως εισηγητής για δύο λεπτά λοιπόν έχετε το λόγο. Εντάξει, αφού μου το ζητάτε θα το κάνω. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για όλες τις ε, ομιλίες γιατί πιστεύω ότι συνέβαλαν τα μάλα στις ε, συζητήσεις μας. Ε, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που προκύπτουν από τις ομιλίες σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την τελευταία παρέμβαση της κυρίας Χαγκητάη. Πολλά καλά μας είπατε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης ίσως ε, θα μπορούσατε να μας πείτε γιατί ε, είναι πλεονέκτημα για σας ε, το ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με το πρόγραμμα FC2. Αλλά να μας πείτε και γιατί δεν βοηθάει και δεν είναι υποφελή συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές τράπεζες. Να μας πείτε ποιο είναι το πλεονέκτημα ε, για την ε, EBRD και το μειονέκτημα για τις Εθνικές Τράπεζες. Γιατί προς το παρόν ζητάμε να υπάρχουν νέα εργαλεία όπως στην Πορτογαλία ακούσαμε ε, ο Πορτογάλος εμπειρογνώμονας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σύστημα τραπεζών, δανειτητικών τραπεζών. Ίσως μπορείτε να μας πείτε και πώς ανταγωνίζεται η μία την άλλη. Αυτό ε, θα μας ενδιέφερε μας. Και κάτι άλλο. Ε, επισημάνατε την περίπτωση την χρήση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το καθεξής. Ίσως ε, τελικά, γιατί για μένα η εντύπωση που έχω είναι ότι δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ε, ναι, μεν υπάρχουν δυνατότητες με το πρόγραμμα ΕΦΣΥ, αλλά ε, δεν υπάρχει πλήρης αποδοτικότητα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ίσως αν όλα αυτά τα συγκεντρώσουμε σε μία ιδέα και μόνο ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο. Γιατί τελικά ε, δεν αποδίδουμε πλήρως. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά επιχειρήματα που αναφέρθηκαν ήδη, αλλά αν εστιάσει κανείς την προσοχή του σε ένα και μόνο θέμα, εσείς τι θα επιλέγατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζουμε με τον εισηγητή της ε, ΕΚΟΝ, Ότμαρ Κάρας, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πολλοί από εμάς ε, στην ανάλυση που έκαναν για τις, και έχουν κάνει κατά για τα υπέρ και τα κατά ε, επιβεβαιώθηκαν σε αυτά που πίστευαν και όλα αυτά καθιστούν απόλυτα σαφές το πόσο σημαντική είναι η αξιολόγηση του προγράμματος FC2. Δεν πρόκειται μόνο για τα περισσότερα χρήματα, ούτε και για το να μπει κανεί σε αυτά τα προγράμματα υψηλού κινδύνου. Εγώ έχω ε, τρεις ερωτήσεις. Κύριε Ζακμάιστερ, εσείς ε, θίξατε το θέμα της ε, ε των ε, counter guarantees για τις επιχειρήσεις. Και θέλω να ρωτήσω, μπορείτε πραγματικά να μας εξηγήσετε το πραγματικό όφελος γιατί υπάρχει κάτι που δεν το έχω καταλάβει καλά. Ε, εμείς ε, ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε στηρίξει αυτές τις επενδυτικές τράπεζες διότι πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν επενδύουν αρκετά στο να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο ε, και ανταυτού τα κράτη-μέλη κάνουν πάρα πολλά για να ενισχύσουν τις επενδυτικές τράπεζες. Εσείς ε, έχετε ίσως ε, κάποια εμπειρία κάτι που να δείχνει από τη δίκη σας στη χώρα ή από κάπου αλλού ότι τα κράτη έχουν στηρίξει περισσότερο τις εθνικές επενδυτικές τράπεζες. Δεύτερο ερώτημα αφορά στη συνεργασία ανάμεσα στις επενδυτικές τράπεζες ε, και τα εγκυοδοτικά ταμεία. Τα επενέσατε αυτά. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε ακριβώς καλύτερα τι πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε οι επενδυτικές τράπεζες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Ο κύριος Μπούλμαν έθιξε ένα θέμα. Υποτίθεται μας ε, μας χαρακτηρίζουν ως διδήμους. Ε, μίλησε για το θέμα της αποτελεσματικότητας της ε, τράπεζας ανασυγκρότησης. Εμείς είχαμε την εντύπωση μέχρι τώρα ότι η Τράπεζα Ανασυγκρότησης δεν κάνει αρκετά για να επιτύχει τους στόχους της. Και εσείς λέτε ότι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο όμως έχει παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Και παράλληλα είναι απαραίτητο να αυξηθεί και το προσωπικό. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ε, στην υποδομή, αλλά ακόμα δεν βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στην Τράπεζα Ανσυγκρότητες και τι πρέπει να γίνει μέσα από το ΕΦΣΥ έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του ΕΦΣΥ. Και άλλη μια τελευταία ερώτηση. Έχετε κάνει εμπειρία με τρίτες χώρες. Ακούω να υπάρχουν όλο και περισσότερα ε, προβλήματα σε σχέση με το Ισραήλ, την Αμερική, ε, με ερευνητικά προγράμματα ε, που εντάσσονται σε προγράμματα συνεργασίες ε, με τρίτες χώρες. Έχετε κάνει κάποια εμπειρία, μπορείτε να μας πείτε τα συμπεράσματά σας. Merci. Σας ευχαριστώ. De la Commission des Budgets. Ο λόγο τώρα στα μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμών. Ο εισηγητή μα, ε, Ζωζέ Μανουέλ Φερνάνδε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για τις ε, ομιλίες τους. Ε, φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης και έχουμε παρόμοιες ε, ανησυχίες. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την προβολή του ΕΦΣΙ, ώστε να γίνει πιο ορατό. Γιατί βοηθήσαμε πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά οι περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν ξέρουν ότι βοηθήθηκαν από ένα ταμείο στρατηγικών επενδύσεων που φέρει τις εγγύσεις του ευρωπαϊκού, του ενωσιακού προϋπολογισμού. Πώς λοιπόν θα βελτιώσουμε αυτή την προβολή. Επίσης, ό,τι φορά τα σχέδια που δεν μπαίνουν καν στο σύστημα. Γιατί εμείς γνωρίζουμε τα σχέδια που είναι στο σύστημα, που εγκρίθηκαν δηλαδή. Τα γνωρίζουμε. Και επίσης γνωρίζουμε ποια προγράμματα ήταν το, το σύστημα, αλλά απορρίφθηκαν. Υπάρχουν όμως κάποια σχέδια που δεν μπαίνουν καν στο σύστημα γιατί τα χαρακτηρίζει πολύ μικρά η ΕΤΕ. Είναι μόνο 25 εκατομμύριο για παράδειγμα, άρα δεν ε, είναι επιλέξιμα για στήριξη. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να μάθουμε ποια σχέδια δεν μπήκαν καν στο σύστημα. Γιατί περισσότερα σχέδια συνδυασμένα ή σε μια πλατφόρμα θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για την υποστήριξη. Επίσης, ό,τι αφορά αυτό το Advisory Hub, τον κόμβο παροχής επενδυτικών συμβουλών, νομίζω και αυτός ο κόμβος μπορεί να συμβάλλει ε, στη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων με την καλύτερη παροχή συμβουλών. Επίσης, ε, μπορεί να προβάλλει καλύτερα το εύση και να βοηθήσει στην αναζήτηση και άλλων λύσεων, στη δημιουργία πλατφορμών για παράδειγμα, προκειμένου να γίνεται ένα συνδυασμό των διαρθρωτικών κονδυλίων με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Για, τις, για τους δημόσιους φορείς είναι δωρεάν η πρόσβαση στον κόμβο επενδυτικών συμβουλών. Και για τι ε, μικρομεσαίε είναι το 1 τρίτο του κόστου. Δεν ξέρω αν οι δημόσιοι φορεί γνωρίζουν ότι είναι δωρεάν η παροχή συμβουλών από τον κόμβο. Το, ο κοινοτικό προπολογισμό αφιερώνει 20 εκατομμύρια το χρόνο σε αυτόν τον κόμβο, κόμβο παροχή επενδυτικών συμβουλών. Αλλά βλέπω ότι οι ανάδοχοι των σχεδίων, οι διαχειριστέ, δεν είναι κανένα τη δυνατότητα αυτή. Πού έγινε το πρόβλημα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα προβάλλουμε καλύτερα αυτό τον κόμβο. Πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό για να γίνει πιο ορατός. Γιατί ε, νομίζω ότι είναι σωστός ο κανονισμός ως προς το στόχο, ως προς το διατακτικό. Αλλά μερικές φορές το πρόβλημα δεν έγκυται στον κανονισμό, στο γράμμα του νόμου, αλλά στην εφαρμογή του. Πώς λοιπόν μπορούμε να τη βελτιώσουμε αυτή την εφαρμογή. Έχετε κάποιες προτάσεις. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Τελευταία. Μιλούμε για την πολυμορφία ή τη μη γεωγραφική συγκέντρωση ή τη μη θεματολογική συγκέντρωση. Θέλουμε μια μεγαλύτερη γεωγραφική και θεματική διασπορά. Ερωτώ λοιπόν, είστε υπέρ ενό στόχου ε, ποσοτικοποιημένου, στο κλίμα για παράδειγμα. Να πούμε ότι για το κλίμα θα πρέπει να έχουμε ένα χι ποσοστό για το κλίμα. Ουσιαστικά κονδύλια ειδικού σκοπού, προσημειωμένα. Θεωρείτε σκόπιμο κάτι τέτοιο. Γιατί η πρόταση για τον κανονισμό προβλέπει ανοιχτή διατύπωση, ανοιχτό κανονισμό, ώστε να εγκρίνονται τα σχέδια που συνάδουν με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ευφύ ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και επίσης να συνάδουν με τις συμφωνίες που έχει συνάψει ή στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σέβεται τη Συμφωνία των Παρισίων, για παράδειγμα, για το κλίμα. Ποια είναι η γνώμη σας ως προς τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε στο κανονισμό ένα ελάχιστο ποσοστό για συγκεκριμένους στόχους, π.χ. το κλίμα. Γιατί ξέρουμε ότι για το ΕΦΣΙ έχουμε φτάσει ως προς τα προγράμματα αυτές στο 40% περίπου η κυρία Γουαρδιασάμπαλ Ρουβιάλ Έφυγε. Τότε να δώσω το λόγο στο συντονιστή μας, τον κύριο Κόλμελ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας ε, για την ε, συμβολή τους και πρέπει να σας πω χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα έχουμε εδώ ε, συγκεντρωμένη τόση πολύ τεχνογνωσία και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας. Ελπίζω να τα κατάλαβα καλά αυτά που μας είπατε και νομίζω ότι με τη δική μου την ανάλυση μας ε, περιγράψατε πάρα πολύ ωραία και με γενικές ε, γραμμές και σε γενικές γραμμές το πόσα ακριβώς μπορεί να είναι ε, θετική όλη αυτή η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως που, μου, που λείπει για μένα είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή. Δηλαδή ε, την έκθεση τη διάβασα λιγάκι και πάρα πολύ ωραία αυτά που μας λέτε και σίγουρα ευσταθούν, όμως θα ήθελα να γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα όσον αφορά τη μόχλευση και τη σορευτικότητα. Τι σημαίνουν ακριβώς όλα αυτά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και εγώ θέλω πραγματικά ε, σε ένα τουλάχιστον ε, πρόγραμμα πρότυπο να μας πείτε πώς ακριβώς υπολογίζετε την προσθετικότητα και τη μόχλευση. Ε, εδώ δουλεύουμε με κάποιες μεσοσταθμικές τιμές που μπορεί να ευσταθούν, όμως θα ήθελα να μας μιλήσετε με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ε, Παραδείγματο χάνει, στη Γερμανία ε, κατασκευάστηκε ένα κομμάτι ενός αυτοκινητοδρόμου και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως ε, επιτυχημένο πρότυπο για άλλα προγράμματα. Έχω λοιπόν μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς, γιατί βεβαίως σήμερα δεν έχουμε και ατελείωτο χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να έρθει κανείς στην ΕΤΕΠ και εσείς ε, να μου διαθέσετε κάποιον ο οποίος για μία ολόκληρη μέρα θα μου εξηγήσει ε, πώς ακριβώς γίνονται οι υπολογισμοί και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν μπορούσατε να μου προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα, πραγματικά αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Τώρα, αν μπορούσατε και τώρα να μου το υποσχεθείτε, θα ήταν και πολύ καλύτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ έτσι το είπα και για αργότερα. Αυτό ήθελα να πω και ίσως μπορεί και κάποιος άλλος συνάδελφος να ρωτήσει κάτι από αυτού. Φυσικά δεν είστε και ο μόνος. Ο κύριος Ρικέ απόν. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι διάκυμε πολύ θετικά προς την εύση. Και αυτό το λέω γιατί ίσως στη συνέχεια ακουστούν επικρίσεις. Στην τελευταία εισήγηση έγινε λόγος για συγκεκριμένα project, προγράμματα όπου ε, η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 95% και το υπόλοιπο 5% ε, αφορά την εύση. Μιλάμε για μία διαδικασία μόχλευσης που δεν συμφέρει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για προσθετικότητα όταν έχουμε τέτοιες ποσοστίες αναλογίες. Αυτό αυτό αφορά και την περίπτωση των 40.000 σπιτιών στη Γαλλία και τη χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Σε μια φάση αποπληθωρισμού θα πρέπει να αρχίσουμε με επενδυτικά σχέδια και να βοηθήσουμε τις χώρες έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα επενδυτικά μέσα για την αντιμετώπιση και του ελλείμματος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεισφέρουμε στη δράση της ΕΦΣΗ. Επειδή ασχολούμε με 15 οδηγίες και κανονισμούς που θα αντικατασταθούν από έναν, θεωρώ ότι και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να προβλέπουν μια σχετική χρηματοδότηση με αυτή της έμφυση, Αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία συνοχής μαζί με το ΕΦΣΥ γιατί δεν συμβαδίζουν τα κριτήρια χρηματοδότησης από τα δύο αυτά ταμεία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η προσθετικότητα, πώς θα υπολογιστεί Πώς υπολογίζουμε το συντελεστή μόχλευσης όταν ε, αναλύουμε την προσθετικότητα. Υπάρχουν επιπρόσθετες ε, επενδύσεις στην οικονομία, γιατί η ΕΕΦΣΗ συγχρηματοδότησε έργα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα γίνονταν, θα προωθούνταν. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές από τους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας υποβάλω τρία ερωτήματα. Κατά την σύλληψη του ΕΦΣΥ πίστευα ότι το ταμείο αυτό θα μπορούσε να ταχθεί υπέρ των υπερεθνικών προγραμμάτων. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι η διαχείριση είναι εθνικού χαρακτήρα και όχι υπερεθνικού. Δυστυχώς. Ο κύριος ε, Κόλμελ μίλησε για την ε, χρηματοδότηση ενός αυτοκινητοδρόμου στη Γερμανία. Γερμανία. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ε, δημόσιες κοινοπραξίες που προβάλλουν έργα που έτσι κι αλλιώς θα είχαν χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, το ΕΦΣΙ δεν είναι ένα μέσο ε, αποσυμφόρησης του, των δημόσιων χρηματοδοτήσεων τη στιγμή που μιλάμε για σύμπραξη δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή στην ουσία το ΕΦΣΙ μετατρέπεται σε ένα μέσο ε, για την αποπαγιοποίηση του δημόσιου τομέα των επενδύσεων δηλαδή και του χρέους πώς συμβάλλει στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη, Δηλαδή, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία δεν θα πραγματώνονταν αν δεν συγχρηματοδοτούσε το ΕΦΣΥ. Τη στιγμή που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς όλες οι συναφείς εγκυοδοσίες από τον δημόσιο τομέα. Γνωρίζετε ε, προγράμματα που δεν θα υλοποιούνταν αν δεν υπήρχε το ΕΦΣΥ. Γιατί στους προϋπολογισμούς ε, έχουμε αυτή την ε, αντίληψη για την προστιθέμενη αξία των ε, ευρωπαϊκών μέσων, δηλαδή το ΕΦΣΥ προσφέρει θέμενη αξία ή είναι ένα επικοινωνιακό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα πρέπει να προωθήσουμε και την απλούστευση. Πιστεύω και εγώ, όπως και εσείς, ότι επειδή θέλουμε να ε, τα καταφέρουμε πολύ καλά, θέτουμε τόσους κανόνες που καταστούν αδύνατη την υλοποίηση των σχεδίων ή τη δυσχεραίνουν. Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές μας, τους εμπειρογνώμονες, θα έπρεπε ίσως να δώσουμε το λόγο και στην ΕΤΕ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. κυρία Καταρίνα Τζαμάρα Ζουτσίντου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να προλάβω την πτήση μου. πρέπει να φύγω. Γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσει την ευκαιρία να απαντήσω τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων πριν φύγω. Μία από τις ε, πολλές ερωτήσεις που άκουσα είναι πώς επιλέγονται τα σχέδια και γιατί, αν λειτουργεί προσθετικότητα, αν έχουν προσθετικότητα αυτά τα σχέδια. Αυτό το ανέφερα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Θέλουμε περισσότερο διαφάνεια για τον τρόπο επιλογής των σχεδίων. Γιατί αυτό που βλέπουμε στον οδηγό είναι ότι τα σχέδια επιλέγονται με βάση τις διαδικασίες του ΕΤΕ, τίποτα άλλο. Και μετά έχουμε ε, διαπραγματεύσεις ε, διμερείς μεταξύ του ε, υποβάλλοντας το σχέδιο ή της πλατφόρμας και της ΕΤΕ. Αλλά δεν είναι και πολύ διαφανής η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την προσθετικότητα, και εδώ προσοχή θα συνιστούσα, γιατί η προσθετικότητα είναι πολύ επίπεδη. Καταρχήν, ένα επίπεδο αφορά την ξεχωριστή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που μπορεί να προέρθει από τα διαρθρωτικά επιδετικά ταμεία, από το συνδέοντα στην Ευρώπη και το καθεξής. Μετά έχουμε ε, προσθετικότητα ανάλογα από το επίπεδο αναγκών του κλάδου. Ε, για παράδειγμα, οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δεδομένη χώρα. Εκεί βλέπουμε τις ροές και υπολογίζουμε την προσθετικότητα. Επίσης έχουμε προσθετικότητα στη δομή του, της του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Εκεί βλέπουμε ότι οι εμπορικές τράπεζες έλεγαν ότι δεν θα δανειοδοτήσουν ένα σχέδιο. Από τη στιγμή όμως που οι βυριδικοί δανεισμοί τύπου μεζανίν ή προέρχονται από την ΕΤΕΙ, το επενδυτικό σχέδιο Γιούγκερ, τότε δέχονται να συγχρηματοδοτήσουν και οι εμπορικές τράπεζες. Αυτή είναι έμπρακτη προσθετικότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν και πολλά στοιχεία της προσθετικότητας σε επίπεδο κινδύνου του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Και εκεί χρειάζονται πολύ πιο αναλυτικές προσεγγίσεις. Αλλά είναι πολυεπίπεδη προσθετικότητα, δεν υπάρχει ένας μονοσήμαντος ορισμός. Επίσης, τι χρειάζεται για να προβληθεί καλύτερα το εύση και να γίνει πιο χρήσιμος ο κόμβος επενδυτικών συμβουλών. Επίσης, ε, ποιο είναι το πιο σημαντικό σύντημα κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Μπούλμαν. Η ευθυγράμμιση είναι το πιο σημαντικό. Τέτοιου είδους σχέδια και τέτοιου είδους πλατφόρμες μπορούν να περάσουν από κάποιες επενδυτικές συμβουλές και χρειάζονται μετά τις συμβουλές ηχή προϋποθέσεις και μετά τις προϋποθέσεις ε, η απόφαση για το αν θα στηριχθεί ε, υποστηριχθεί το σχέδιο. Θα πρέπει σε όλες αυτές τις φάσεις να υπάρχει προβολή και ορατότητα. Επίση, ό,τι αφορά την ικανότητα, το δυναμικό. Αν μιλούμε για ανθρώπινο δυναμικό, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Όταν ξεκινήσαμε το 2007 το πρώτο χρηματοοικονομικό και χρηματοδοτικό μέσο, δεν είχαμε αρκετό προσωπικό. Και όταν μιλούμε για δυναμικό, ε, ενώ δυναμικό ως προς τις γνώσεις, δηλαδή η ΕΤΕ έχει πολύ περισσότερες γνώσεις για το πώς αντιμετωπίσει διάφορα είδη κινδύνων. Και αυτό που προβάλλεται είναι ότι αυτό που προτείνουν τις περισσότερες φορές είναι μέγεθος μόνο, όγκος, αλλά αυτό δεν αρκεί. Υπάρχουν περισσότερα πράγματα και έχει την τεχνογνωσία η ΕΤΕ, αλλά χρειάζεται και προσωπικό και ανθρώπινο δυναμικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, προσημείωση για κάποια κονδύλια θα μπορούσαμε στην εξάντε αξιολόγηση αναχώρα που έγινε, που έγινε πριν το 2014 είπαμε ότι υπήρχαν κάποια κονδύλια προσημειωμένα για τα ευρωπαϊκά και διαρθρωτικά, ε, επενδυτικά και διαρθρωτικά κονδύλια. Και εκεί μπορούμε να δούμε τις συγκεκριμένες ανάγκες ε, σε μια χώρα για κάθε τομέα. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλές εκπομπές για παράδειγμα, αλλά οι χώρες είναι πολύ διαφορετικές, ε, οπότε δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε υπερεθνικό στόχο για την προσημείωση. Καλύτερα να δούμε ε, τι χρειάζεται σε κάθε χώρα περισσότερο για να πούμε περισσότερα κονδύλια να αφιερώσουμε στις μεταφορές ή περισσότερα στην ενέργεια, ανάλογα όμως με τις θετικές ανάγκες κάθε χώρας και κάθε τομέα, όχι σε διακρατικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Δεν θα δώσω λοιπόν το λόγο ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε στο Συμβούλιο, γιατί στις 7 τη Δευτέρα το απόγευμα θα συνεδριάσουμε στο Στρασβούργο. Δευτέρα το απόγευμα θα έχουμε σχετική συνεδρία στο Στρασβούργο και εκεί θα μιλήσουμε και για το ΕΦΣΙ και για το ΕΦΣΙ 2. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει, ο κύριος Σέκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ετέθησαν. Έγιναν κάποιες ε, γενικής φύσεως ε, παρατηρήσεις. Θα αναφερθώ και εγώ σε κάποιες γενικές και πιο ειδικές ε, παρατηρήσεις δικές μου. Όσον αφορά το πρόγραμμα ΕΦΣΥ, το πιο βασικό ερώτημα ετέθη στο τέλος το κάνατε εσείς. Δηλαδή κάποια προγράμματα δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ε, χωρίς το πρόγραμμα ΕΨΗ. Στην κατάσταση ως έχει τώρα όπου υπάρχει επαρκής ρευστότητα και χαμηλά επιτόκια, αν υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα με μεγάλη κερδοφορία, ε, δεν θα πάει κανείς, δεν θα στραφεί στο ΕΦΣΥ, διότι θα βρει τη λύση στην αγορά. Το βασικό λοιπόν στοιχείο του ΕΦΣΥ έχει σχέση με την κερδοφορία των προγραμμάτων ε, το οποίο εξορισμού η κερδοφορία αυτή είναι χαμηλότερη από ότι η αγορά ε, θα στήριζε υπό φυσιολογικές συνθήκες και το άλλο, το σημαντικό, είναι η ποιότητα των προγραμμάτων. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι το θέμα της αποδοτικότητας είναι πολύ σημαντικό και το πρόγραμμα ΕΦΣΥ μέσα από το μηχανισμό του είναι σε θέση να αυξήσει την αποδοτικότητα της κερδοφορίας. Εγώ ε, σας μίλησα για την πρόσμιξη, το διαγωνισμό αυτό ε, που δημοσιεύτηκε σήμερα για μεταφορές και υποδομές μεταφορών. Εδώ έχουμε μια πολύ καλή περίπτωση. Η κερδοφορία αυτού του προγράμματος ε, θα μπορούσε να συνδυαστεί με το πακέτο χρηματοδότησης, άρα δηλαδή κάτω στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Όμως ε, όταν πρωτοεμφανίστηκε το πρόγραμμα ΕΦΣ ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς ε, περί σε πρόκειτο. Οι περισσότεροι που στηρίζουν τέτοιου είδους ε, προγράμματα ε, παρενέβησαν και έτσι η ποιότητα του προγράμματος ε, δεν ήταν πάντα προσαρμοσμένη σε αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ιδιωτικός μηχανισμός με δημόσια εγγύηση, όπως είναι το ΕΦΣΥ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνει κάποια αξιολόγηση, δηλαδή ποια προγράμματα ε, θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί χωρίς το ΕΦΣΥ, ίσως η πλειοψηφία ε, στις ε, μεταφορές και στην κοινωνία τα περισσότερα δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί αλλά θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ ε, που το θέμα αυτό του κόμβου των, ε, της παροχής συμβουλών ε, το ότι συζητήθηκε το θέμα αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καλούμεθα να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση. Ε, βεβαίως αυτή είναι μια δική μου παραδοχή, αλλά θα εξακολουθήσει να ασκεί κατά την άποψή μου στο μέλλον, γιατί θα υπάρξει έλλειψη κονδυλίων. Τώρα, όσον αφορά τα ε, διασυνοριακά προγράμματα, στις μεταφορές με το ΕΦΣΥ δεν μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει μια σύραγγα, αλλά μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποια κομμάτια του προγράμματος τα οποία συμβάλλουν στην επιτυχία του διασυνοριακού προγράμματος. Ε, συμφωνώ μαζί σας, ε, αυτή είναι μια δυναμία, πρέπει να συνεχίσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά τελικά νομίζω ότι ε, κάτι μπορούμε να πετύχουμε. Και τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να θίξω ένα θέμα, δηλαδή σε κάποιες προηγούμενες παρεμβάσεις έγινε λόγος ε, για την επίδραση των ΣΔΙΤ σε δημοσιονομικές απαιτήσεις. Από τη μια δηλαδή προσφέρει κανείς κονδύλια και από την άλλη αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Εμείς στη Γενική Διεύθυνση MOVE και με την βοήθεια συναδέλφων και άλλων γενικών ε, διευθύνσεων ε, νομίζω κάνουμε μια πολύ χρήσιμη δουλειά με τη Eurostat και ε, συμπεριλήφθηκε και η ΕΤΕΠ τέλη Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε ένας οδηγός για την στατιστική αντιμετώπιση των ΣΔΙΤ στο δικό μας τομέα. Ίσως να είμαι πολύ αισιόδοξο. Αλλά αυτό μπορεί να εκλειφθεί ως ένα σημείο εκκίνησης για να εξετάσουμε και άλλου είδους θέματα για να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Και πραγματικά συστήνω ανεπιφύλακτα με βάση αυτή την πολύ καλή αρχική επίδοση συστήνω οι εργασίες να συνεχιστούν και σε άλλες εξίσου σημαντικές κατευθύνσεις. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά ο κύριος Ζωζέ Φερνάντο Φιγκέιρέδο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις θα προσπαθήσω να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο-τρεις πτυχές που ε, αφορούν δικές μου αρμοδιότητες. Στο, στην αρχική σας δήλωση υπήρξε μία πρόταση κατά πόσο χρειαζόμαστε, δηλαδή χρειαζόμενοι καλύτερες ε, επενδύσεις, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Βεβαίως, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε σχέση με τον επιμερισμό επενδύσεων του ΕΦΣΥ. Και εδώ δεν μιλώ για μία κοινοπραξία και το πώς ε, την χάνει διαχείριση, τι διαχείριση την χάνει, αλλά θα πρέπει να αποτιμήσουμε τα χαρτοφυλάκια όταν ε, φτάνουν στον αρμόδιο φορέα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ε, περιθώρια μόχλευσης, άρα υπάρχει και δυνατότητα χρησιμοποίησης της αξιολόγησης του τριπλού α και έχει μεγάλη σημασία το ποια διαδικασία αξιολόγησης ακολουθούν γιατί δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Όλα τα βλέπουμε ε, σε σχέση με τον κίνδυνο, τα επίπεδα κινδύνου και τον επιμερισμό του. Εάν μιλάμε για καινοτόμα σχέδια ή νεοσύστατες εταιρείε, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση, ε, εάν υπάρχει σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικού τομέα, να υπάρχει μεγαλύτερη ροή χρήματος όταν πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο, ας πούμε. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την περιφερειακή ανάπτυξη των αναδόχων, διότι αν αναλύσουμε μία πρόταση που προέρχεται από τη μεσημβρινή Ιταλία ή από το κέντρο του Παρισιού ή του Βερολίνου, η απάντηση δεν είναι η ίδια. Και στη μία περίπτωση θα υπάρξει έγκριση, στην άλλη απόρριψη. Δεν λέω ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο αυτό το κριτήριο, γιατί διαφορετικά θα χαθεί το τριπλό α. Και ως υπεύθυνο υπεύθυνος για τα χρηματοδοτικά θα πρέπει να σας τονίσω τη σημασία και τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια πρόσμιξης χωρίς να αλλάξει η συνολική διαδικασία διότι από ό,τι κατάλαβα από ε, μία ε, παρουσίαση που έγινε από το ΕΦΣΙ και από το ε, Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει πάντα σωστή ε, προσέγγιση γιατί προσπαθούν να αποκτήσουν χρήματα σε χαμηλή τιμή. Κάτι το οποίο προαπαιτεί ένα τριπλό αλφα. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε εμείς ότι μπορείτε να αποκτήσετε χρήμα και λίγο ακριβότερα αν χρειαστεί, αλλά σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις της αγοράς. Το δεύτερο θέμα αφορά την προσθετικότητα και τα κριτήρια αποτίμησης της αποτελεσματικότητας του Ταμείου. Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο για την αξιολόγηση, αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων, όχι μόνο με βάση την προσθετικότητα, αλλά και με δύο-τρία άλλα κριτήρια. Η προσθετικότητα είναι σημαντική, αλλά επίσης όταν μιλώ για προσθετικότητα, μιλώ για ε, τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα που είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο αλλά έχει σημασία και η αποτελεσματικότητα των μέσων. στο φάσμα των δικτών θα πρέπει να εμπεριέχεται και αυτό. Δηλαδή, να, ε, αυτό που έχει σημασία είναι η προσθετικότητα, δηλαδή περισσότερα χρήματα στον ανάδοχο, αλλά η ουσία είναι κατά πόσο επιτυγχάνουμε το στόχο μας. Γι' αυτό θα περιλάβω και ορισμένα άλλα κριτήρια και σε κάποιο άλλο στάδιο των εργασιών μας θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, σε σχέση με το γεωγραφικό καταμερισμό και τις πλατφόρμες, μπορώ να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία όχι μόνο προς την, ως προς την παρούσα χρηματοδότηση, αλλά και σε άλλα επενδυτικά πλαίσια. Όταν μιλάμε για τέτοιες δομές, μπορούμε να έχουμε πανευρωπαϊκές δομές. Αν έχουμε όμως μικρές επιχειρήσεις και εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν είναι εύκολη η σύσταση μιας τέτοιας πλατφόρμας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό γιατί υπάρχουν και νομικές, ρυθμιστικές και φορολογικές δεσμεύσεις. Όταν προβαίνουμε στη σύσταση μιας πλατφόρμας για επενδύσεις στο Σαν Φρανσίσκο, ξέρουμε ότι θα υπάρχει το ίδιο χρηματοπιστωτικό και φορολογικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Αμερική. Στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ο οργανισμός που εκπροσωπώ σήμερα, ο πορτογαλικός αυτός ο οργανισμός, ε, ασχολείται με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και, στη και τη διαχείρισή τους στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Άρα, για να γίνει το σχήμα λειτουργικό δεν πρέπει να δούμε μόνο το χρηματοπιστωτικό πακέτο, αλλά να προχωρήσουμε και στη σύσταση ορισμένων ε, τμήματων των ευρωπαϊκών αγορών. Διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μία λύση που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ε, καταστάσεις και τη ζήτηση. Δηλαδή, αν γίνει σύσταση μίας ε, πλατφόρμας στην Αυστρία, και θέλω να κάνω μία επένδυση σε μία πορτογαλική εταιρεία και εδώ και κάτι το εναλλακτικό στη Γερμανία, ίσως η κατάσταση να είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τη γραφειοκρατία και τον εταιρικό φόρο από ότι αν, κάνω, αν προβώ στη σύσταση αυτής της πλατφόρμας στο Παρίσι, στη Μαδρίτη ή στο Βίλνιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Τέλος. ο κύριος ε, Ούντο Μπούλμαν μίλησε για το γεγονός ότι η απόδοσή μας είναι χαμηλότερη από το προσδοκόμενο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι αυτά τα μέσα, επειδή είναι πολύ χρήσιμα και γι' αυτό τα ανέφερα στην παρουσίασή μου, και θα ήθελα επ' να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, αυξάνουν τον προϋπολογισμό αν δούμε τις ε, καινοτόμες εταιρείες και την καινοτόμο εργασία ως προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι βάζουμε χρήμα στο, στην αγορά, αλλά τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν όπως θέλουμε, αν ε, δεν λάβουμε υπόψη και την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή τις πληροφορίες, και τη ζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο σε σχέση με τους στόχους. Γι' αυτό οι συμβουλευτικές ε, πλατφόρμες μπορούν να βοηθήσουν έναν επιχειρηματία έτσι ώστε το εύση να μην το δούμε μόνο από την πλευρά της ζήτησης. Αυτό είναι το ευκολότερο αλλά το δυσκολότερο είναι να υπάρχει και η πραγματική προσφορά την οποία επιθυμούμε. Και έτσι θα μπει χρήμα και στις, στις οικονομίες μας και στις χώρες μας για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Όταν λέτε ότι η ΕΤΕ ε, ανησυχεί για το τριπλό της α, αυτό σημαίνει ε, ότι επειδή θέλει να κρατήσει το τριπλό α δεν αναλαμβάνει πολλούς κινδύνους και γι' αυτό ε, βρίσκεται κάτω των προσδοκιών ενός εύση. Κάτι το οποίο δεν αναλαμβάνει, δηλαδή κινδύνους που δεν αναλαμβάνει η αγορά. Η ξεκάθαρη μου απάντηση είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ισχύει αυτό που λέτε, είναι καταθετική απάντηση, όχι παντού, γιατί πολλά σχέδια είναι δημόσια, αλλά ένα τμήμα της αγοράς μπορεί να προσκρούσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά για τις δημόσιες συμβάσεις δεν έχετε πρόβλημα, έχουν κρατική εγγύηση. Ναι, αλλά για τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις γιατί δεν, έχουν, δεν υπάρχουν εγγύσεις. Ναι, αλλά για τις δημόσιες συμβάσεις ε, δίνονται κρατικέ εγγύσει, οπότε δεν έχουν πρόβλημα οι αγορές. Αλλού είναι που έχουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μπερνάρ Σάγκμαϊστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να απαντήσω κυρίως ε, στον Ευρωβουλευτή κύριο Κάρας, δηλαδή ποιο είναι το πραγματικό όφελος. Και θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο παράδειγμα της Αυστριακής Τράπεζας Επενδύσεων. Το ΕΦΣΙ λοιπόν οδηγεί στο ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε περισσότερους κινδύνους και επίσης μπορούμε να παρακολουθήσουμε περιπτώσεις με χαμηλή φερεγγιότητα. Εδώ προκύπτει η προσθετικότητα. Βεβαίως αυτά δεν μπορούμε να τα ποσοτικοποιήσουμε γιατί εξαρτώνται από τη ζήτηση και η ζήτηση κυμαίνεται. Το θέμα είναι όμως ότι όχι μόνο μπορούμε να αναλάβουμε περισσότερους κινδύνους, αλλά με το πρόγραμμα που έχουμε, το επενδυτικό, μπορούμε να εφαρμόσουμε και περισσότερα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Ε, τώρα πάω στο δεύτερο ερώτημα. Τι είδους προσπάθειες ε, καταβάλουν τα κράτη-μέλη για να συμβάλλουν. Ε, και πάλι θα σας αναφέρω το παράδειγμα της Αυστρίας. Δηλαδή χρειαστήκαμε κάποιο χρόνο μέχρι πολιτικά να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά. Αλλά εντωμεταξύ είμαστε σε μια περίοδο όπου ο προπολογισμό μας αυξάνεται κατά 50% σε σχέση με παλαιότερα. Υπάρχει λοιπόν και άλλη μια ε, προέκταση του ΕΦΣΙ, προκύψει από το ΕΦΣΙ, ότι μπορούμε να λάβουμε περισσότερους κινδύνους και έτσι λοιπόν, και ίσως με αυτόν τον τρόπο απαντάτε και η προσθετικότητα, στην ε, περίπτωση της Αυστρίας, στην εξάντε αξιολόγηση των προγραμμάτων, εξετάζουμε επακριβώς μακροοικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή ένα πρόγραμμα, πόση καινοτομία να έχει, η ανάπτυξη θα προκύψει. Και αν οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε περισσότερους κινδύνους. Με ένα και μόνο πρόγραμμα έχουμε, αναλαμβάνουμε περισσότερους κινδύνους ή δεχόμετα μία επιχείρηση η οποία ε, λειτουργεί με χειρότερους όρους. Κατόπιν το θέμα ε, των ε, κοινοτικών θεσμών. Εγώ αυτό θα το θυμάστε, το προέβαλα και είπα ότι έχουμε τον, τη δική μας την ένωση, την Ένωση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εγκυοδοσίας. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τα μέλη μας. Ε, και έτσι έχουμε συγκεντρώσει τις γνώσεις μας και μπορούμε αυτές να τις ε, μεταφέρουμε στους ε, θεσμούς. Ε, γιατί όσον αφορά τα μέλη μας, σημαντικότερες βέβαια είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς συμμετέχουμε άμεσα στην αγορά, γνωρίζουμε πολύ καλά τις αναγκαιότητες και έτσι λοιπόν ε, οποτεδήποτε εφαρμόζονται νέα προγράμματα μπορούμε να παρέμβουμε. Και πάλι στην Αυστρία, στην πιλωτική φάση, στο Ινοφίν, είχαμε για τα δικά μας τα προγράμματα ένα πολύ μικρό πιλωτικό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε απλά ε, έχοντας κατά νου να δούμε αν, θα, αν είναι λογικός ο σχεδιασμός. Και διαπιστώσαμε ότι η τιμολόγηση δεν ήταν επαρκής. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το στοιχείο, ε, το στοιχείο αυτό λήφθη υπόψη από τους ε, σχεδιαστές, προέβησαν στις απαραίτητες αλλαγές, άρα καταλαβαίνετε ότι όλη η συνεργασία είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σουζάνα Χαρκιτάη, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν αποφασίσαμε τη θέσπιση του ΕΦΣΙ, και αναθέσαμε τη διαχείρισή του στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εσείς στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δεν διαρωτηθήκατε γιατί δεν λάβατε και εσείς μέρος αυτή τη διαχείριση, γιατί 72% της ΕΤΑ ανήκει σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά χρειάζεται και εσείς να περάσετε μέσω της ΕΤΕ. Δεν διαρωτηθήκατε λοιπόν γιατί εσείς δεν λάβατε μέρος όπως και οι ΕΤΕ στη διαχείριση. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω πρώτα σε δύο-τρία άλλα ζητήματα και είμαστε στη διάθεσή σας και για περαιτέρω θέματα και απαντήσεις. Καταρχήν, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε πιο στενά με το ΕΦΣΥ ε, σας είπα ότι εμείς έχουμε την όρεξη του κινδύνου, μας αρέσει ο κίνδυνος και εξετάζουμε το θέμα του εμπορικού κινδύνου όταν χρηματοδοτούμε σχέδια. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα. Λίγες ε, εταιρείε στην ε, στις περιφέρειες που ε, δραστηριοποιούμαστε χρειάζονται κάποια επιχειρησιακή αναδιάρθρωση των οικονομικών τους. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και συνήθως δεν το αναλαμβάνουν άλλοι συνάδελφοι. Γιατί λοιπόν στην Ελλάδα, στην Ρωμανία, στην Κροατία δεν ε, μπορούμε να συνεργαστούμε με τις άλλες τράπεζες ε, για να μοιραστούμε τον κίνδυνο και να προβούμε στην αναδιάρθρωση. Εμείς χρειαζόμαστε κάποιον που παραλαμβάνει περισσότερο κίνδυνο. Και φαίνεται ότι μεταξύ του 2008 και του 2010 και μετά είχαμε και την κρίση, οπότε είχαμε πολύ λίγες εταιρείες που ενδιαφέρονταν. Επίσης, Έχουμε μια περιφερειακή σιδηροδρομική επιχείρηση. Χρειάστηκε νέο τροχαίο υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, καλύτερες υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως ε, τα συμβόλαια δημοσίων κρατικών προμηθειών ήταν οχθέτους διάρκειας, ενώ η χρηματοδότηση θα προϋπάθεται 15 ετή ορίζοντα και δεν μπορούμε να ε, χορηγήσουμε αν δεν έχουμε σύμβαση δημοσία σύμβαση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από κοινού, με κάποια διαβρύση του κινδύνου. Ναι, φυσικά χρειάζονται, θα έχουμε καλύτερε υπηρεσίε, δεν χρειάζονται καν διαρθρωτικά ταμεία, δεν χρειάζονται καν κρατικέ εγγύσει, αλλά λίγο ένα επιπλέον ποσοστό κινδύνου που θα πρέπει να αναλυφθεί από κάποιον άλλον, γιατί όχι από το ΕΦΣΥ. Επίσης έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία ε, παροχής ενεργειακών υπηρεσιών που λαμβάνει ε, συμβόλαια από διάφορους δήμους. Χρειάζεται λίγο μετοχικό κεφάλαιο. Εμείς μπορούμε να αναβάνουμε ένα τμήμα, αλλά θέλουμε και έναν άλλο να επομιστεί το υπόλοιπο τμήμα του κινδύνου. Έχουμε λοιπόν τέτοιου είδου σχέδια που θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε συνεργασία, να αναπτύξουμε πλατφόρμες και σε αυτό το συμπλήρωμα που χρειαζόμαστε θα μπορούσε εκεί να μπει η ΕΦΣΗ. Επίσης, εταιρείε που χρειάζονται κάποια οικονομική αναδιάρθρωση για να κάνουν περισσότερες επενδύσεις. Έχουμε πολλές τέτοιες. Και αυτές οι εταιρείε χρειάζονται λίγο επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο, λίγη αναβάθμιση και εμείς χρειαζόμαστε ένα εταίρο για να μοιραστούμε τον κίνδυνο. Τώρα, γιατί δεν συνεργαζόμαστε με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Εσείς μας ζητήσατε να συνεργαστούμε με ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες. Αυτή είναι η εντολή μας, να προωθήσουμε τις εμπορικές επενδύσεις. Οπότε οθούμε τις εμπορικές τράπεζες που είναι εταίροι μας να ξεφύγουν λίγο από το χώρο που αισθάνονται άνετα για να συνεργαστούν μαζί μας, για να μην το παίζουν μόνο εκ του ασφαλούς. Επίσης, θέλουμε να μετακινούμαστε γιατί συνεργαζόμαστε μαζί τους σε παράλληλη χρηματοδότηση στην περιοχή που ενεργοποιούμαστε εμείς από τη Βαρσοβία μέχρι την Αθήνα Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Εκεί έχουμε αναπτυξιακέ τράπεζε που έχουν τη δυνατότητα και το δυναμικό να χρηματοδοτήσουν κάποιες, ε, κάποιο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό με εμά. Αυτό είναι, το θέμα είναι η εντολή μας περιορίζει και επίσης δεν είναι τυχαίο που σε μερικές χώρες έχουν ε, ξεχωριστά τα ταμεία στη σχέση με τις αναπτυξιακές τράπεζες. Άλλος, κάνει την αναπτυξία άλλος, άλλες είναι οι δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Τράπεζας, άλλος κάνει το Financial Engineering. Επίσης, στις χώρες, 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε μεγάλη κάλυψη γεωγραφική. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε το ΕΦΣΥ. Επίσης και στο κόμβο ε, χρειάζεται κάποια αποκέντρωση. Εμείς έχουμε τέτοια αποκέντρωση, φτάνουμε σε, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στους ε, αναδόχους των ε, σχεδίων και για μεγαλύτερα σχέδια υποδομών, για δημόσιες υπηρεσίες, για εταιρείε μέσης κεφαλαιοποίησης, καλό θα είναι να έχουμε άμεση επαφή και αυτή την αποκέντρωση την εξασφαλίζουμε εμείς. Γιατί δεν μπορούμε το εύση να το περάσουμε από, το, από τις τραπεζικές ενέργειες μέσω διαδικτύου. θέλουμε προσωπική επαφή, θέλουμε να φτάνουμε στις εταιρείε αυτές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τα mid-caps. Σε ό,τι αφορά τη μόχλευση, μπορώ και εκεί να σας αναπτύξω πολλά επιμεροσημεία, γιατί εσείς ε, μας πιέζετε και κάθε φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να τους κάνω ένα τεστ αγοράς για να τους πω αν υπάρχει μόχλευση ή αν στριμώχνω τους ε, εμπορικούς μας Και το θέμα είναι τι μου φέρνετε κάθε φορά διαφορετικό με ρωτάνε σε σχέση από τα απλά, τον απλό τύπο σχεδίων. Και τα τελευταία 20 χρόνια κάθε σχέδιο περνάει από τέτοιο εξονυχιστικό έλεγχο. Και το, συνδυα... το συζητώμε και στην ε, ΕΤΑ και οι, οι πολιτικοί θέλουν προσετικότητα και κλίμακα. Για να φτάσουμε σε οικονομίες κλίμακος θέλουμε συσσόρευση και μεγαλύτερη εστίαση στην προσετικότητα. Γιατί οι προσδοκίες είναι πολλές και για τη μόχλευση ε, και γι' αυτό θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες και πραγματικά νιώθουμε αλληλέγγυοι προς την ΕΤΕ που μέσα ε, σε πολύ λίγο χρόνο χρειάστηκε να, ε, να δείξουν τέτοια αποτελέσματα και ως προς την προστατικότητα γιατί ήταν υψηλότητα της προσδοκίες και πραγματικά ήταν σημαντικό το έργο τους. Σας ευχαριστώ. Τώρα ε, οι εισηγητές μας για τη δεύτερη φάση του ΕΦΣΥ θέλουν το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ζωζέ Μανώλη Φερνάντες. Εντάχει απλώς να σας ευχαριστήσω οι παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που έχουμε ως προς το ΕΦΣΥ. Λειτουργεί καλά, άρα μπορούμε να το βελτιώσουμε το Ταμείο αυτό Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό απορρέει από τη συζήτηση. Από τη δική μας πλευρά θα θέλαμε το FC2 να ε, είναι ένας κανονισμός που να είναι έτοιμος μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ελπίζω το Συμβούλιο να είναι στο ύψος των περιστάσεων και αυτού του στόχου. Το θέμα της προσθετικότητας είναι ένα ε, θέμα ουσίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τον ορισμό της ναι, ναι, ναι. προσθετικότητας. Θεωρώ ότι καταρχήν υπάρχει ο στόχος και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θέλει να προωθήσει τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σαφές. Θα συνεχίσουμε με τη συνεισφορά των εμπειρογνωμόνων που έκαναν εξαιρετικές εισηγήσει. Το εύση που εντάσσεται στο σχέδιο Juncker είναι ύψη της σημασίας για την Ευρώπη. Είναι ένα μικρό παιδί, πολύ απαιτητικό αυτή τη στιγμή ε, δεν έχει κλείσει τα δύο του χρόνια, αλλά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Αντίθετα με αυτό που πίστευαν πολλοί που αμφισβητούσαν τη σημασία αυτού του ταμείου για όλα τα κράτη-μέλη ε, απαιτεί ε, ενεργές παρεμβάσεις από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Γίνονται επικρίσεις προς την ΕΤΕ και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά η ΕΤΕ άλλαξε. Με βάση το ΕΦΣΥ πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα και επιβάλλεται διάβια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την έγκριση ενός προγράμματος ή την απόρριψή του. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους εμπειρογνώμονες για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε. Ούντο Μπούλμαν. Λοιπόν, και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονες ε, και όλους τους υπόλοιπους. Πραγματικά έμαθα πάρα πολλά, πρόεδρε και συμπρόεδρε. Και θα τα συνοψίσω. Θα τα πω ε, για να ξέρουμε και τι θα κάνουμε στα στις επόμενες φάσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ε, πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος ε, με αυτή την προσέγγιση ε, γιατί νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα ΕΦΣΙ αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Να είμαστε αποτελεσματικοί για τι περιοχές, για εκείνου που χρειάζονται επιπρόσθετε ποιοτικέ επενδύσεις και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το διγονήμα για μα και στο νομοθετικό κομμάτι. Αυτά όλα συμβαδίζουν και με την άποψη που είπε η Καρτατσίνα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως ε, το δυναμικό καινοτομίες που υπάρχει βέβαια στην Τράπεζα Ανασυγκρότησης αλλά και σε άλλους ε, θεσμούς. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Φιγκερέντο ο οποίος είπε ότι ε, υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα σε ένα ταμείο που λειτουργεί με μόχλευση και πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα 3α αφενός αυτό και από την άλλη και ο πολιτικός στόχος που συνοδεύει το ΕΦΣΥ που είναι να αναλαμβάνει αναλαμβάνονται περισσότεροι κίνδυνοι. Υπάρχει δηλαδή ε, κάποια αντίφαση ανάμεσα από τα δύο. Εγώ να πω το εξή. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις. Γιατί όταν μιλάμε για ΕΤΕΠ, εμείς είμαστε οι βασικοί φορείς της ιδέας. Και όπως είπε και ο Χωσέ, να αλλάξω το χαρακτήρα μου, να αλλάξω το προφίλ μου και μετά να επανέλθω στα κανονικά απλά με τη δικαιολογία ότι η προπόθεση είναι τα 3α, ε, αυτό δεν γίνεται, δεν βοηθάει καθόλου. Ε, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες άλλες δυνατότητες. Και ο κύριος ε, Ζάκμαρ μας είπε με ποιες δυνατότητες μπορούμε να κάνουμε εξάντε αξιολογήσεις και να καταλήγουμε σε ένα μεικτό χαρτοφυλάκιο που να λέει αυτή είναι η κατάσταση και θα πρέπει ε, να αναλάβετε περισσότερους κινδύνους για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν για να μείνει κανείς στην αγορά. Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε από την τράπεζα ανασυγκρότησης είναι ότι ε, θα είναι απόλυτα διαφανής ε, με τέτοιου είδους προβλήματα. Συμφωνώ επίσης ε, ότι υπάρχουν και δυνάμει αντιφάσεις ανάμεσα στην ποιότητα και τον όγκο, την ποσότητα. Πρέπει να είμαστε πολύ ε, επιφυλακτικοί από αυτού και ίσως ε, σε περαιτέρω νομοθετικές πράξεις να αποφασίσουμε από αυτού. Αν θέλουμε το ΕΦΣΙ να είναι η πρώτη δυνατότητα επενδύσεων στην αγορά, τότε θα πρέπει εξάντε εκ των προτέρων να ορίζουμε τις επιπτώσεις και την ποσότητα, τον όγκο. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επίσης ε, θα πρέπει και πολιτικά να νομιμοποιήσουμε ε, και το προφίλ αυτό ότι το ΕΦΣΙ είναι πρωτοπόρος στις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ τους παρεμβαίνοντες εμπειρογνώμονες για τις πολύτιμες γνώσεις τους. Ευχαριστώ τους εισηγητές και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που ήταν άκρος διαφωτιστική. Φιλοδοξούμε ώστε το εύση και το, ιδιαίτερα το εύση 2 να είναι ένα ειδικό μέσο που να καταδείξει ότι χωρίς αυτό οι επενδύσεις δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Και πώς να αναλαμβάνουμε έναν κίνδυνο τη στιγμή που δεν τον αναλαμβάνει η αγορά. Χρειάζεται απλούστευση, γιατί εάν υπάρχει απλούστευση θα είναι και η επικοινωνία πολύ καλύτερη και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σύγκληση των νομοθεσιών και των εθνικών ρυθμίσεων. Μία από τις μεγαλύτερες τροχοπέδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτός ο κατακαιρματισμός του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Πρέπει να ε, προοδεύσουμε και ήδη βλέπουμε ότι το ευρώ και η ευρωζώνη γίνονται πιο ε, εύρωστες και επίσης θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά, τα επενδυτικά κενά που υπάρχουν και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους συμπροέδρους. Κάτι ίσως έχει να πει ο κύριος Γκουαλτιέρη, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι εισηγητές και με τα συμπερασματικά του σχόλια μπορούμε να συνοψίσουμε με τρία στοιχεία. Προσθετικότητα που δεν είναι μια γραφειοκρατική ετικέτα, είναι μια συνεχής προσπάθεια για επιπρόσθετες επενδύσεις ε, με βάση την ποιότητα και την αντιμετώπιση των ελλείψεων της αγοράς καθώς και καλύτερη νομοθέτηση και ενίσχυση της νομοθεσίας σε σχέση με τις συνήξεις που θα πρέπει να γίνουν, η χρήση των εθνικών πλατφορμών και ούτω καθεξής. Και φυσικά χρειάζεται ενεργή συμμετοχή, όπως είπε ο κύριος Φερνάντες. Ενεργή συμμετοχή των θεσμικών οργάνων και της ΕΤΕ. Και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συνεισφέρει σε αυτή την ενεργό συμμετοχή. Και φυσικά χρειάζεται καλύτερη, μεγαλύτερη διαφάνεια για να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις όχι μόνο στην νομοθεσία αλλά και στην διαχείριση. Ε, Δυστυχώς, μάλλον το εύση είναι ένα μικρό παιδί, το οποίο όμως θα μεγαλώσει και θα μας βοηθήσει στην διαχείριση και διακυβέρνηση του εργασιακού πλαισίου στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτό το πολύ χρήσιμο σεμινάριο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πριν συνοψίσουμε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το τμήμα ε, θεματικών ενωτήτων και ιδιαίτερα τον κύριο Πέρτινς, ο οποίος ε, ειδικά εκείνος μας βοήθησε ε, ιδιαίτερα για τη συγκρότηση αυτού του τμήματος.